Okay, good morning everybody. Good morning. Καλημέρα σας συνάδελφοι. Καλημέρα και στο κρατήριό μας από το διαδίκτυο, γιατί η συνεδρίασή μας μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Καλημέρα σε όλους σας λοιπόν. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να προσθέσω και δύο σημεία αν δεν έχετε αντίρρηση. Την ψηφοφορία για την έκβαση του τριμερούς διαλόγου για το πακέτο ε, για τα ταξιδιωτικά και επίσης ε, το 68 ε, για το εξοπλισμό πίεσης ε, από το Συμβούλιο της 15 Απριλίου και επίσης το σημείο 9 την ιστορία που αναποδοχικά από, τα οδικά οχήματα και το σημείο 10 για, για τα, τις νέες Προκλήσει ε, από τον τουρισμό που θα γίνει αντιστροφή των δύο σημείων στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αλλαγέ, παρακαλώ να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Περνάμε στις ανακοινώσει τη Προέδρου. Καταρχήν η αντιπροσωπή μα στο Λουξεμβούργο. Ακυρώθηκε η επίσκεψη στο Λουξεμβούργο γιατί δεν ε, υπέβαλαν ε, αρκετά μέλη οι πολιτικές ομάδες για συμμετοχή στην αντιπροσωπεία. Και επίση θα ήθελα να σας ενθαρρύνω όσο προχωρούμε προς την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μορφή για τη συνεδριάση, το e-meeting, να λαμβάνετε τα έγγραφα από εκεί, για να πρωτοστατήσουμε εμεί την ψηφιακή αγορά. Τώρα, ενημέρωση για τις, τους τριμερείς διαλόγους. Α, προηγουμένω τα πρακτικά αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη 23η Απριλίου. Εντάξει. Περνάμε στην ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους. Βλέπω την Κάθριν ε, για τους εξοπλισμούς για τα καλώδια, ε, τις με αέριο. Καταρχήν, Κάθριν. Δεν έχω να σα πω και πολλά. Έγινε η πρώτη συνεδρίαση για τις συσκευέ με αέριο. Ένα θέμα έχουμε με την ενίσχυση για το μονοξίδιο, το άνθρακα. Στον επόμενο τριμερή διάλογο θα εξετάσουμε τη θέση του Συμβουλίου. Ήταν πολύ παραγωγική και καρποφόρη συνεργασία. Φαίνεται ήταν δεκτικό το Συμβούλιο. Δεν έχουμε πολλές διαφορές, αλλά για το θέμα αυτό του μονοξιδίου του άνθρακα θέλουμε ε, μια ισχυρή διατύπωση, γιατί είχαμε την είδηση για τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τη διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Οπότε θέλουμε τέτοιες συσκευές με αέριο να είναι ασφαλείς και να έχουν ανοιχνευτές ε, για να ανοιχνεύουν αμέσως οποιαδήποτε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Το θέμα αυτό είναι απολύτως ε, απαραίτητο να ληφθεί υπόψη είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια των πολιτών. Θα επανέλθω μετά, την επόμενο, μετά τον επόμενο τριμέρι διάλογο. Μάλιστα. Καταρχήν έχετε σχόλια για αυτό, για τους τριμερείς διαλόγους, είτε για τις συσκευές με αέριο, είτε ε, το άλλο με τα καλώδια. Δεν είμαι εγώ η εισηγήτρια για τις άλλες εκθέσεις. Ε, Καταρχήν για τα διακοσμητικά αγάντια για το φούρνο και για το πλήσιμο των πιάτων. Εμείς θέλουμε να το αποκλείσουμε, το Συμβούλιο να το συμπεριλάβει. Είναι προσυζήτηση το θέμα. Η πρόεδρος μας είναι η συγγήτρια. Τώρα για τα καλωδιακά. Βλέπω κάποιους και οδησηγητές που παρακολουθούν το θέμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος να μας ενημερώσει. Νομίζω έχουμε τον εισηγητή. Είναι πιο αρμόδιος για να μας ενημερώσει. Περιμένω πάντως ε, τις διαπραγματεύσεις και για το προστατευτικό εξοπλισμό και για τις συσκευές με το αέριο. Βλέπω τον κύριο Λόπες Ιστουρής. Μήπως μπορεί να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις από τη ε... Σας ευχαριστώ. colegas, eh, en el ámbito del, del informe sobre sistemas. Σε ό,τι αφορά το, τα συστήματα μεταφορά με καλώδια τελεφέρι κλπ. Ε, από τι 182 τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιτροπής ε, διαπραγματευθήκαμε το Συμβούλιο καταφέραμε να βελτιώσουμε την αρχική πρόταση. Έχουμε τέσσερα σημεία στα οποία μένουμε στις τροπολογίες. Η μία αναφέρεται στην ιστοσελίδα, δεύτερο στο σύστημα πέδησης, σε αυτά τα συστήματα μεταφοράς τελεφερικ μέσω καλωδίων και τρίτο θέμα, την αρχή της προφύλαξης, precautionary principle. Το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα έστειλε τις νέες συμβαστικές τροπολογίες και προτάσεις και θέλουμε να παραμείνει μνήμα στο website, στην ιστοσελίδα που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια νέα διατύπωση για τα συστήματα πέδησης, για να κρατήσουμε την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητα, ένα πληρέστερο άρθρο για το σύστημα των κυρώσεων και επίσης αγκαταλείψαμε ε, την τροπολογία που αφορά την αρχή της προφύλαξης, γιατί υπάρχει στις άλλες ε, εξαίσθηση ε, ευθυγράμμισης για τις συσκευέ με αέριο και τους του προστατευτικούς ε, μηχανισμούς. Και πιστεύω ότι στις 11 Ιουνίου θα γίνει ουσιαστικά ο καταληκτικός τριμερής διάλογος της χειραψίας που λέμε για να ολοκληρώσουμε την διαπραγμάτευση γιατί έχει προχωρήσει πολύ τεχνικά το θέμα, είναι αίσια η έκβαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και την Πρόεδρο, τη Βίκη Φόρτ, που συνέβαλε τα μάλα για τη σύναψη τη συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο και πάλι στην Κάτριν Σίλερ να μας ενημερώσει τι γίνεται για την ομάδα εργασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Θέλετε να πείτε κάτι για τις ε, συσκευές με καλώδια, για τις εγκαταστάσεις αυτές. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την υποστήριξή του για τα θέματα που ανέφερε, τα οποία είναι ακόμα σε συμβιβασμό, αλλά έχουν προχωρήσει πολύ. Και ιδιαίτερω η επιτροπή μα αυτή είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για το θέμα των κυρώσεων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει των ε, προστήμων. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Και όσοι έχουν τα πράγματα σήμερα, έχουμε μια πιο ε, αυστηρή ρήτρα και στο διδακτικό και στις ιδεολογικές σκέψεις. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το υπογραμμίσω. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο, κυρία Άντρουσον. Κάποιο άλλο σχόλιο από πλευρά των μελών για του τριμερεί διαλόγου. Πολύ ωραία. Προχωράμε λοιπόν τώρα στην ενημέρωση από πλευρά τη κυρία Στήλερ για την ομάδα εργασία για τα δικαιώματα διανοητική ε, ιδιοκτησία και πνευματική ιδιοκτησία και για τη μεταρρύθμιση. Κάνετε μια συνεδρίαση το Μάιο. Σα ευχαριστώ. Δύο συνεδριάσει στι 13 και στι 28 Μαου. Στις 13 Μαΐου έγινε μια ενημέρωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλυση για την δημοσίευση και από πλευρά των εμπλεκομένων φορέων θέματα έθεσαν για τα πνευματικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά τον τομέα της μουσικής. Είναι πολύ ωφέλιμη αυτή η δελαγή απόψεων. Οι προτάσεις έγιναν το φθινόπωρο και ήταν χρήσιμε και νομίζω ότι το γεγονό ότι συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορεί ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά η συνεδρίαση του Μαΐου ήταν καλή. Έγινε μία μελέτη από το Κέντρο για τις Ευρωπαϊκές Μελέτες για τα θέματα αυτά Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη και η παρουσίασή της. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για την Επιτροπή μας να την μοιράσουμε. Γιατί πέρα από ότι ήταν συναρπαστική, μας δίνει μια καλή εικόνα του τι συμβαίνει σε άλλα κράτη-μέλη, την διαφορετική εικόνα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Μία από τις τελευταίες συζητήσεις επικεντρώθηκε στο πώς διασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία θα αντέξει στο μέλλον σε βάθος χρόνου. Και τονίστηκε ότι η νομοθεσία θα ενημερωθεί. Αλλά αν θέλουμε να επιλύσουμε κάποια από τα ζητήματα που έχουμε, μπορούμε να το πράξουμε ήδη από τώρα. Και τι βλέπουμε στην ψηφιακή πραγματικότητα. Δεν είμαι και ειδική σε θέματα ξέρετε. Μπορούμε όμως έτσι να προασπίσουμε την νομοθεσία με την κωδικοποίηση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις ε, κρύβεται αλγόριθμοι πίσω από αυτά. Και νομίζω λοιπόν ότι χρήσιμο θα ήταν να ενημερωθούμε και για αυτή την ακαδημαϊκή πτυχή. Μάλιστα, λέει η πρόεδρο, υπάρχει κάποιο άλλο μέλο τη ομάδα εργασία για τα πνευματικά δικαιώματα που θα θέλει να πάρει το λόγο να σχολιάσει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα σα ε, μοιράσουμε την ε, έκθεση αυτή. Καλή ιδέα. Μάλιστα, να ξεκινήσουμε λοιπόν στις 9 και μίση την ψηφοφορία Προβλέπετε τουλάχιστον και 9.30, αλλά ας μην ξεκινήσουμε πιο νωρίς γιατί ίσως έρθουν και άλλοι, και άλλοι συνάδελφοι. Άρα ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 9.30. Uh, dear colleagues, let's start with the vote. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε όλοι μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας, τις ηλεκτρονικές, γιατί θα ξεκινήσουμε. Κάθριν, εσύ. Yes, okay. Uh, okay, uh, I would like to say that some of the colleagues of the EPP are not... Θέλω να πω ότι κάποιοι συναδέλφοι από το ΕΛΚ δεν βρίσκονται εδώ, γιατί έχουμε τη συνάντηση του Προεδρείου του Βουδαπέστη. και έτσι η συγγητρία κυρία Γκάλπελτ δεν βρίσκεται εδώ, θα την αντικαταστήσει ο κύριος Σάνφελ. Θα θέλετε να πείτε κάτι ε, για το σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά τον προπολογισμό 2016 και την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Όχι, οπότε προχωράμε στην ψηφοφορία. Amendment 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Παρακαλώ συναδελφοί, ας ξεκινήσουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2, καταπίπτει. 3, υπέρ, 2. πρέπει να την ψηφίσουμε, υπέρ, κατά,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 αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 πρώτο τμήμα έχουμε ψηφοφορία τα τμήματα εδώ πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τελική ψηφοφορία για το σύνολο της ε, γνωμοδότησης με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν άπαντες. We count you as well. Ωραία, υπολογίζουμε και εσάς συν, ζητώ συγγνώμη, μία ε, παραπάνω ψήφους από το άλλο. Συναδελφοί, πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη, διότι είχαμε μία ψήφο παραπάνω από ό,τι έπρεπε από το Άλντε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν ανάπαντες Ψηφίζουμε υπέρ. Ωραία. Πέρα ψηφοφορία. εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Yeah, uh, colleagues, now we have to uh, vote to actually. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια ψηφοφορία έγκριση ουσιαστικά προκαταρκτική πρόταση πιλωτικών έργων ή ε, παρασκευαστικών δράσεων προπαρασκευαστικών πράξεων. Θεωρούμε ότι εγκρίνεται το σχέδιο αυτογνωμοδότηση καθώ και των πολιτικών σχέδιων και προπαρασκευαστικών πράξεων εγκρίνεται. Okay, colleagues, now we vote on Mr. Boussoy report να ψηφίσουμε την έκθεση του για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, τροποποιητικό κανονισμό 107-2009 για την εμπορία προϊόντων φωτιά. Τροπολογία. Ατιμή. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κάτα. Αποχές. Έλεγχο παρακαλώ. Για την 30 παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, απορρίπτεται, διορθώνει ο Πρόεδρος. Συμβιβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική μάλλον τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ίντα 9. Με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ε, είχαμε ετοίμα για ονομαστική κλίση από τους πράσινους, αλλά δεν επαρκεί ο ρυθμός των μελών, άρα δεν θα είναι ονομαστική κλίση. Είναι τα εννέα υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε έναν έλεγχο. Είναι τα εννέα. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Και εσείς ε, υπέρ. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε στη 36. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Η 37. Είναι ταυτόσιμη, δεν την ψηφίζουμε. Η 38, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν στην συμβαστική παριθμών 4. Πρόκειται για ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Και τώρα. Συμβαστική τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 14 συνάδελφοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και περνάμε στις συλλογικές σκέψεις. Τροπολογία 10. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 11. Α, είναι όλα ταυτόσιμες. Άρα περνάμε στη 14. Στη 13, συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όλες καταπληκτούν Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι δύο. Η τρία της ίντα. Υπέρ, κατά, αποχές. Θέλετε να ελέγξουμε. Μάλιστα, έναρξη ψηφοφορίας για την ίντα 3. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. ψηφίσατε όλοι για την 3. Α, περισσεύει μία ψήφος από το ΕΛΚ. Υπεράριθμη μία ψήφος. Θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε. Ποιος ε, λοιπόν ψηφίζει και δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Ξανά λοιπόν συνάδελφοι από την αρχή. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφορίας για την ΙΝΤΑ 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Γιατί έχουμε και δύο συναδέλφους οι οποίοι ψηφίζουν χωρίς κάρτα. Περνάμε στην τροπολογία υπερθμών 20. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Όλοι τα υπόλοιπα καταπίπτουν και έτσι λοιπόν περνάμε στην τροπολογία 28. Α, έχουμε και μία ακόμη της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου, είναι τα πέντε, λοιπόν. Είναι τα πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Δύο ψήφοι λείπουν. Λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η ψηφοφορία. We congratulate. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Κρίστιαν Μουσόη. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την εντολή ε, για την έναρξη τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο. Πρέπει να γίνει ονομαστικά, με ονομαστική κλίση για την ε, για την εμπορία προϊόντων φώκες, έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο Εντολή. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Οπότε εγκρίνεται η εντολή για τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Ωραία, θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την σύσταση προγράμματος ε, για λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις ε, και πολίτες, διαλειτουργικότητα ως μέσο εξυγχρονισμού του δημόσιου τομέα. Μήπως θέλει η κυρία Γιακοσάρη, η να λάβει το λόγο. Όχι, απλώς να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις ηγητές για την πολύ επικοδομητική συνεργασία. Ελπίζω από το πρόγραμμα αυτό να υποφεληθούν ε, κυρίως οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Συμβεστική τροπολογία 3. 3ε. Ποιος είναι υπέρ. Η Ρόζα. Ε. Ποιος είναι υπέρ. Συμβαστική τροπολογία ε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 76. Τα αντίστοιχα τμήματα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 84. Οι υπόλοιπε είναι γλωσσικές. 83. Ποιος είναι υπέρ. 83. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ξεχάσαμε την 80... 82, 83, 82, 84 83 είναι παρομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Περνάμε στην τροπολογία 87. Ποιος είναι υπέρ. 85 διορθώνει η πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ. Το F το κάναμε, το ψηφίσαμε. 85. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 86. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 87. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία G. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 90. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 λέει η πρόεδρος. 18. Α, σίγουρα τα γυαλιά μου τα χρειάζομαι, οπωσδήποτε. 18 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 18. Τροπολογία 97. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Αντίστοιχο τμήμα ένα τμήμα 1. Ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. τροπολογία 100, το 3, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 102, καταπίπτει. Τροπολογία 103. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία K. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία 111. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 117, αντίστοιχο 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία L, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 119. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία M. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 37. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 126. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 128 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. 46 λίβρος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την τροπολογία 1. Amendment 1. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Ρούζες. I close the vote and it is adopted. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται η τροπολογία 1. Τροπολογία 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 51 αντίστοιχο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία. Συμβαστική τροπολογία C. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική τροπολογία Δέλτα. Δι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοπαλία 17 προς 17, άρα απορρίπτεται. Τροπολογική 63. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 65 παρακαλώ, άρχεται ψηφοφορία voting with is developing. Do I have the it's yours voting? I close the vote. Τέλος. Απορρίπτεται. Now an oral amendment on a... Προφορική τροπολογία τώρα επί της 66 τροπολογίας. Ρούζα Τούν. Να τη διαβάσω. Ή δεν χρειάζεται. Όπως θέλετε, από εσάς εξαρτάται. Δεν χρειάζεται, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν δεν θέλετε να τη διαβάσετε, ας την ψηφίσουμε κατευθείαν. 66 με την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 και 69 που είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 απο, έχει αποσυρθεί 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σας ευχαριστώ συνάδελφοι τελική ψηφοφορία τώρα ήταν πολύ υπομονετική πάντως, μπράβο σας. Με ονομαστική κλίση, ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότης. Άρχεται η ψηφοφορία. The driving economy. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια κυρία Γιακονσάρη αδελφοί, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση Ταραμπέλα προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα. Θα ήθελε ο εισηγητής να πει δυο λόγια. Όχι. Κύριε Ταραμπέλα, θα θέλετε να πείτε δυο λόγια. Δεν θέλω να καθυστερήσω την ψηφοφορία, κυρία Πρόεδρε αλλά θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης που συμμετείχαν στις δύο συνεδριάσεις ε, μελέτης και διαπραγμάτευσης των τροπολογιών. Η δουλειά έγινε με πολύ, καλό, πολύ καλή ατμόσφαιρα και συνεργασία και ελπίζω να παραλυφθεί το ίδιο και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Συναδέλφοι, συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά δεν ψηφίζει κανένας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική 3 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ε, τροπολογία 20. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, Συμβεβαστική 5. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 21, την τροπολογία 21. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες, πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Συμβεβαστική 5 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την τροπολογία 25 ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Στα, ε, στις σκέψεις, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές ε, κρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την έκθεση Τάρα Μπέλα προς μια ακμάσουσα οικονομία που ε, βασίζεται στα δεδομένα ψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον κύριο Σιγητή. we also have Συνάδελφοι, πρέπει επίσης να εγκρίνουμε ένα προφορικό ερώτημα που σχετίζεται με την έκθεση Ταραμπέλα. Μπορούμε να την εγκρίνουμε. Ωραία, λοιπόν, θα θεωρήσουμε την προφορική ερώτηση. Εγκρίνεται. Colleagues, we are We have not finished the votes yet. Αδελφοί, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα την ψηφοφορία. Πρέπει να ψηφίσουμε για την ε, έναρξη των τριμερών διαλόγων για τα οργανωμένα ταξίδια και τις διευθετήσεις ε, ε, για τα ταξίδια με συνοδεία και Μπρίγκετ Λάγκε θέλετε να πείτε κάτι. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδης και την ομάδα που μας περιέβαλε. Οι διαπραγματεύσει ήταν αρκετά δύσκολες. Στις 5 Μαΐου επιτύχαμε πολιτική συμφωνία και 28 Μαΐου το Συμβουλίο Ανταγωνιστικότητα υιοθέτησε το κείμενο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, όπως επίσης και το ότι τα δύσκολα σημεία ήταν δυνατόν να υιοθετηθούν και η προστασία των καταναλωτών στο σύνολό τη έχει ενισχυθεί. Οι καταναλωτές τα καταλαβαίνουν καλύτερα τα δικαιώματά τους ως αποτέλεσμα. Είναι ε, καλά όλα αυτά που πετύχαμε. Θα δούμε σε τρία χρόνια κατά πόσο λειτουργούν και φέρνουν αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας να εκδηλώσετε ε, τη συμφωνία σας. Ε, κύριε Κιάμπερτ, έχετε το λόγο. Εξ ονόματι της ομάδας μου ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγητρία για τη δουλειά της. Πράγματι το θέμα αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για τη δική μας ομάδα. Απογοητευτήκαμε λίγο από το αποτέλεσμα, όχι γιατί δεν δουλέψα αρκετά, αλλά διότι ε, το θέμα που μας απασχολεί είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι αυτό που μπλόκαρε το ζήτημα αυτό. Και πιστεύω αυτό ε, το θέμα, οι υπουργοί να εμποδίζουν να επιτύχουμε καλύτερα δικαιώματα για τους καταναλωτές είναι κάτι αρνητικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά καλά πράγματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν βάσει της έκθεσης, οπότε παρά όλα τα προβλήματα η ομάδα μου θα υποστηρίξει τη γνωμοδότηση και σε τρία χρόνια θα επανεξετάσουμε την κατάσταση και εκείνη τη στιγμή θα δούμε τι έχει συμβεί και εκεί θα μπορέσουμε να δώσουμε την τελική μας συμφωνία. Αλλά θα πρέπει να αποδώσουμε και ευθύνες σε όσους εμπόδισαν την επίτευξη καλύτερων δικαιωμάτων για τους καταναλωτές. Ευχαριστούμε, εκτιμάμε ιδιαίτερα, την ευελιξία που δείχνετε. Άρχεται η ψηφοφορία, συνάδελφοι, για την υιοθέτηση της έκφρασης ε, των τριμερών διαλόγων ε, για ε, τα οργανωμένα ταξίδια και τα ταξίδια με συνοδεία. ξύψαν άπαντες. Θα θεωρήσουμε λοιπόν ότι η έκφραση του τριμερούς διαλόγου έχει εγκριθεί. Τελική ψηφοφορία τώρα για τις νομοθετικές πράξεις και τα άλλα μέσα, το corrigendum, το διορθωτικό αυτό διορθώνει την οδηγία 2014-68 για την εναρμόνιση των νόμων των κρατών μελών που σχετίζονται με διέθεση στην αγορά εξοπλισμού πίεσης που είχε υιοθετηθεί ήδη στην προηγούμενη θητεία. Πρέπει να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. I open the vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Από όσο βλέπω το διορθωτικό εγκρίνεται. Thank you very much everybody. And now we... Ευχαριστώ άπαντες και περνάμε τώρα στη συζήτηση με τη γνωμοδότηση για τις νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη. Συντάκτρια είναι η κυρία Γκραπίνη και σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Κυρία Γκραπίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Am pregătit un proiect de aviz din partea INCO pentru, destinat Comisie pentru Transport și Turism. Λοιπόν, προσπάθησα να προετοιμάσω αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για την INCO, αλλά δεν ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί εγώ είμαι μέλος και των δύο επιτροπών αλλά θεωρώ ότι εντός της ΙΜΚΟ θέλουμε να βρούμε νέες έννοιες για την πρόθεση του τουρισμού, ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησα στο σχέδιο αυτογνωμοδότησης να αποδείξω σε ποιο βαθμό είναι σημαντικός ο τουρισμός για την Ευρώπη, για την εσωτερική αγορά. Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι γιγάντιες και ε, μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εμείς ε, λέμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την ανάπτυξη του τουρισμού και η ψηφιακή πλατφόρμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τουρισμό είναι εξαιρετική, ε, σημαντική για να βοηθήσει να δώσει περισσότερες δυνατότητες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και νέες πλατφόρμες ε, τις οποίες δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει και επινοήσει ε, οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένω να βοηθήσουν την Ευρώπη να βελτιώσει ε, την ποιότητα και την ποσότητα των πληροφοριών που δυνανται να βρουν οι καταναλωτές. Η ΙΜΚΟ πιστεύω θα πρέπει να υπογραμμίσει την πτυχή αυτή. Χρειάζονται καλύτερε διαπραγματεύσει και συνέργειες μεταξύ χωρών στον τομέα του τουρισμού στο νου μου έχω λέγοντας αυτό τους επισκέπτες από την Κίνα, από την Ινδία, από την Κορέα οι, οποία, οι οποίοι ε, θα μπορούσαν να αγοράσουν ένα ταξίδι που, με το οποίο θα μεταβαίνουν σε πολλές ε, διαφορετικές χώρες με μια ενιαία τιμή. Ε, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατών ώστε να μπορούμε να προτείνουμε ένα ταξίδι τέτοιου τύπου ε, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ε, επαληθεύσιμες και ελπίζω ότι θα λάβουμε από όλες τις πολιτικές ομάδες κάποιες προτάσεις. Εγώ προσωπικά έχω ακόμα τροπολογίες να προτείνω και θεωρώ ότι όσον αφορά την ΙΜΚΟ ε, η ΙΜΚΟ μπορεί να προσφέρει κάποιες καλές ιδέες στην Επιτροπή Μεταφορών διότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμα εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον, στον κύριο Κοέγιο του του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μα την κυρία Γραπίνη για το σχέδιο που υπέβαλε και να πω ότι συμφωνώ μαζί τη σε ό,τι αφορά την εκτίμηση που έκανε του τουριστικού κλάδου γιατί πραγματικά είναι σημαντικό μοχλός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τουρισμό. Και έχουμε επίγνωση ότι ο τουρισμός είναι ένας σημαντικό οικονομικός κλάδος και είμαστε ο πρώτος ε, τουριστικός προορισμός. 9% του ΑΕΠ παγκοσμίως σχετίζεται με τον τουρισμό και είναι και επίση σημαντικό τομέα δημιουργίας θέσεων απασχόληση. 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ε, έχουν κάποια θέση εργασίας ε, που σχετίζεται με τον τουρισμό. Οπότε είναι ένα ζήτημα που έχει άμεση σχέση με τους καταναλωτές, όπως είπε και η συγκεκριά κυρία Γκραπίνη. Και δεδομένης της ε, τεχνολογικής εξέλιξης έχουμε άθηση και του τουρισμού και μάλιστα μέσω όχι παραδοσιακών διάβλων, πολλοί, όλοι και περισσότεροι πολίτες κάνουν τις κρατήσεις τους ε, μέσω του διαδικτύου. Οπότε κάπου συμπίπτει το νέο ψηφιακό θεματολόγιο με την ανάπτυξη και τις εξελίξεις στον τουρισμό. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ψηφιακή διατησία στα θέματα του τουρισμού. Τι θα αποφαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια νέα διάσταση που διαμορφώνεται με τις νέες τεχνολογίες. Και το θέμα της προστασίας του καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και ε, μια και η δική μας Επιτροπή είναι η Επιστοπή Προστασίας του Καταναλωτή, είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στις όλες τις ζητήσεις. Επίσης, έχουμε το ευαίσθητο και λεπτό θέμα των ευάλωτων καταναλωτών. Γιατί με τη γύρεση του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι κάνουν τουρισμό. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς τους πιο ευάλωτους καταναλωτές ε, για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να μπορούν να τα απολαμβάνουν απρόσκοπτα. Στα πλαίσια της έκθεσης ε, Γκραπίνη θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε το πολύ σημαντικό θέμα. Το ΕΛΚ θα καταθέσει και τροπολογίες και ελπίζω να συνεχιστεί η καρποφόρα συνεργασία μας ώστε η γνωμοδότηση της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ να είναι χρήσιμη για την αρμόδια καθήλια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Μεταφορών και να βελτιωθεί πραγματικά το εύρος και το περιεχόμενο της έκθεσης της Επιτροπής Μεταφορών. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο, εκ μέρους των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, ο κύριος Ντάλτον. Um, Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρους του ECR αλλά και του Ρίτσαρτ Σέλοκ που είναι ο Σκιώδης που δυστυχώς δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει. Έχουμε συμμετήσει καλή εντύπωση για αυτό το σύνδεο γνωμοδότηση. Δύο σχόλια από πλευρά μα, πάντα έχουμε δύο σχόλια. Αλλά όχι πολύ κακά. Το ερώτημα στην παραγραφό 4, αυτή την πρόταση του να υπάρχουν ευρωπαϊκοί χάρτες ε, ταξιδιών ε, στην εφαρμογή online. Η ερώτησή μας είναι πώς θα το χρηματοδοτήσουμε αυτό. Ε, αυτή η χρηματοδότηση θα προσθέσει αξία. Ένα μικρό ερώτημα λοιπόν γι' αυτό. Όταν δεν υπάρχουν πολλά χρήματα όπως αυτές τις εποχές πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις χρηματοδότησης και μετά ο κ. ήθελε να θέσει το σημείο για τα θεωρήσεις και τη φορολογική σε ορισμένα ζητήματα. Ειδικότερα το ζήτημα φορολογική είναι θέμα επικουρικότητας. Οπότε μας ανησυχεί η συμπεριλήψη της ε, φορολογίας στην παραγραφό 5. Θέλουμε να αφαιρεθεί διότι θεωρούμε ότι είναι θέμα κρατών μελών. Ε, είναι, αυτά είναι τα κυρία σχόλια του κ. Σολέκα. Εγώ ως ε, πολίτης του ξέρετε μας... Ε, οι, οι, οι θεωρήσεις της ζώνης δεν μας αφορούν άμεσα, αλλά έμεσα. Γιατί ξέρετε, οι κανόνε που χρησιμοποιεί για τη ζώνη Σέγγεν η Ευρώπη μα έχουν επιπτώσει και σε εμά. Πρέπει δηλαδή όταν αλλάζουν αυτοί οι κανόνε να κάνουμε κάτι κι εμεί. Οι δικοί μα κανόνε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για την Κίνα για παράδειγμα, είναι πιο ευέλικτοι από ότι στην ε, ζώνη Σέγγεν. Αυτό είναι μια παρατηρήση μου. Και η τρίτη μου, το τρίτο μου σχόλιο. Εγώ είμαι στην Task Force για τον τουρισμό στην Επιτροπή Μεταφορών και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να προωθήσουμε για την ανάπτυξη του ε, τουρισμού είναι να μειώσουμε τα τέλη των αεροδρομίων για να ενθαρρύνουμε την έλευση τουριστών στην Ευρώπη, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε, όταν πετάει στι Βρυξέλλε, στο αεροδρόμιο των Βρυξελών και δει στο εισιτήριο τι φόρο πληρώνει για να πετάξει προ και από το αεροδρόμιο των Βρυξελών, αυτό ε, δεν βοηθά τον τουρισμό. Κάνει την Ευρώπη πολύ πιο ακριβή, ε, υψηλή φόρη των αεροδρομίων στην Ευρώπη κάνει την Ευρώπη λιγότερο ελκυστική. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό σε εθνικό επίπεδο, να ε, ασκήσουμε κάποια πίεση για τη μείωση των φόρων αεροδρομίων, διότι ε, αποτελούν πρόσκομα για την οικονομική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στη για την ΑΛΔΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Γραπίνη έκανε έργο πολύ καλή ποιότητα που θα μα ε, χρησιμεύσει ω ε, βάση. Ε, συμφωνούμε για τι ευκαιρίε του τουρισμού. Θα ήθελα μόνο να πω. Να πούμε ότι πρόκειται για την ανάπτυξη όλου του πλανήτη. Δεν πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να θεωρεί ότι έχει πλεονέκτημα. Πρόκειται για ανταγωνισμό. Και νομίζω λοιπόν ότι πρέπει ο τομέας αυτός να χαρακτηριστεί από πιο έντονο επαγγελματισμό, να υπάρχει, ε, υπάρχει καλή ποιότητα και καλά επίπεδο σε όλα τα, κατα... σε όλα μελη Σε ό,τι αφορά όμως συγκεκριμένα την ΙΜΚΟ, θα ήθελα να εκφράσω δύο στοιχεία και δύο απόψεις σε ό,τι αφορά και τις προτάσεις για τροπολογίες. Η πρώτη σε ό,τι αφορά τα θέματα τα ψηφιακά. Έχουμε την πρόοδο τη ψηφιακή τεχνολογία στον ταυτό τομέα και πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε σχέση με τον καταναλωτή. Δύο παρατηρήσει ήθελα να κάνω. Θα σα παρουσιάσω τη λογική. Ήδη έχουμε κινητοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πλατφόρμες ε, κάπως ηγεμονικές όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους πολίτες και στους καταναλωτές. Αυτό αληθεύει και στον τομέα του τουρισμού. Ξέρετε, ορισμένε αμερικάνικε πλατφόρμε για τι οποίε έχουμε συζητήσει πολύ τι τελευταίε εβδομάδε ε, έχουν αναπτύξει τουριστικέ δραστηριότητε. Άλλε είναι γνωστέ ω παγκόσμιοι ηγέτε ε, στο ξενοδοχειακό τομέα και πρέπει η Ευρώπη να ε, έχει τα μάτια ανοιχτά, διότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμό, πρέπει να υπάρχει πλουραλισμό, όχι να υπάρχει μόνο μία πλατφόρμα. Και εδώ αναφέρομαι σε ιδιωτικέ πλατφόρμε, ιδιωτικέ τοποθεσίε δεν ε, αναφέρομαι στην πλατφόρμα της Κομισιόν για, που προωθεί το τουρισμό. Θεωρούμε, θεωρούμε ότι ο τουρισμός πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα όσα λέμε εμείς για τον πλουραλισμό, από την ανταγωνιστικότητα. Το δεύτερο, γνωρίζουμε όλοι ότι οι τουριστικές πρακτικές σήμερα υπογείται στην έλευση νέων πρακτικών που αποτελούν προκλήσεις. Ας δούμε το Airbnb, το Uber. Συνεργατικές πρακτικές είναι αυτές στον τομέα του τουρισμού. Άνθρωποι που νοικιάζουν ε, διαμερίσματα δικά τους ιδιώτες. Ε, όλες αυτές οι πτυχές του τουρισμού έχουν ανοίξει ξαφνικά ε, παράλληλα με το επαγγελματικό, με το επαγγελματικό κομμάτι του τουρισμού. Ε, και αλλάζουν τις πρακτικές που υπάρχουν. Εγώ δεν έχω κάποια ένσταση με όλα αυτά, αλλά θέτουν προκλήσεις. Οπότε στο κειμένο πρέπει να προσθέσουμε αυτές τις προκλήσεις που εμφανίζονται, διότι παρότι θέλουμε να εκφραστεί, να υπάρχει δημιουργικότητα, πρέπει παράλληλα να προστατεύουμε τα δικαιώματα των όσων να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες σε ιδιώτες ε, και να προστατεύουμε και τα δικαιώματα των ε, ε, τουριστών επίσης. Ε, είναι θέμα αριθμιστικό. Το έχουμε κάνει σε πολλούς άλλους τομείς και πρέπει να το τονίσουμε και στον τομέα του τουρισμού. Ε, πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε πολύ αποτελεσματικά για όλα αυτά. Ευχαριστούμε κύριο Ροσφόρ. Δίνω τώρα το λόγο ε, για τους πράσινους του κύριο Σωτές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Γραπίνη για την ε, γνωμοτότηση αυτή. Όλοι συμφωνούμε ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κλάδο στην Ευρώπη. Και ότι στο μέλλον πολλά θα είναι τα έσοδα τα οποία αναμένουμε από τον κλάδο του τουρισμού. Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλέον ανταγωνιστικούς σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία και ασφαλώς επηρεάζει και άλλους πολλούς τομείς. που με τη σειρά του συμβάλλουν στον τουρισμό. Να διευκρινίσω ότι συμφωνώ με την κυρία Κραπίνη σε ό,τι αφορά την ανάγκη επένδυση στον τομέα του τουρισμού προκειμένου να υπάρχουν και ε, εξελίξεις ε, στον κλάδο. Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται οι απειλούμενες ε, ομάδες. Σε ό,τι αφορά τώρα τους, τα ταξίδια πακέτο, που συμπεριλαμβάνουν δηλαδή ε, όλες τις πτυχές του ταξιδιού. Θα πρέπει στον τουρισμό να προστατεύονται όλοι οι καταναλωτές. Και νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί στα πλαίσια του τρομερού διαλόγου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον... Ε, και το Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε την προστασία του καταναλωτή σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η πρόεδρο. Δεν βλέπω να ζητάει κανένα άλλο το λόγο από πλευρά του EFD. Άρα το λόγο λοιπόν τώρα έχουν τα μέλη τη Επιτροπή. Ο κ. Δαντιέ, έτσι το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Μαρία Γραπίνη για την καταπληκτική τη γνωμοδότηση. Είναι κάπω περίεργο ότι η τρίτη οικονομική κοινωνικονομική δραστηριότητα της Ένωσης ό,τι αφορά τη συμβολή στο ΑΕΠΑ και τη συμβολή στην απασχόληση είναι και είναι από τους τομείς που συνεχίζουν να αναπτύσσονται παρά την κρίση και παρόλα αυτά είναι σχετικά άγνωστος τομέας για τα θεσμικά όργανα. Πιστεύω ότι τα θεσμικά όργανα θα έπρεπε κυρίως να ασχοληθούν με αυτό το τομέα που είναι πολύ σημαντικός. Πριν από λίγο μάλιστα εγκρίναμε μια πολύ σημαντική συμφωνία με το Συμβούλιο για, το τουριστικό, για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τα τουριστικά πακέτα. Θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε την αξία που αξίζει σε αυτό το, σε αυτό τον κλάδο, σε αυτή την κατηγορία. Επίσης ε, έχουμε πολύ σημαντικά πολιτιστικά ατού και γεωγραφικά, ιδηλιακά τοπία και μέσα από του σημαντικότερου παγκοσμίου ε, προορισμού. Επίση, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ψηφιακή εποχή για να έχουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει σημαντικό κατακαιρματισμό και πολύ φραγμή. Επίση, η ταξινόμηση των ξενοδοχείων. Ε, είναι πολύ διαφορετικά τα αισθήματα ταξινόμηση των ξενοδοχείων στην Ευρώπη. Κατακαιρματισμός λοιπόν. Ενώ η παγκόσμια τουριστική αγορά είναι όλο και πιο ανταγωνιστική και αυτή την άποψη θα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα στον τουρισμό. Γι' αυτό και οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουν και θα πρέπει να αξιοποιήσουν στον τουριστικό κλάδο. Και έχω και μία, υπενθυμίσω μία πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα ευρωπαϊκό σήμα τουριστικής ποιότητας. Βέβαια προς το παρόν είναι προαιτικό αυτό το σήμα, αλλά θα μπορούσε να δώσει ακόμη μεγαλύτερη προβολή στα συστήματα, τα τουριστικά μας. Και κυρίως ε, το θέμα της υποδοχής και της φιλοξενίας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας ε, λέει η συγγήτρια της γνωμοδότησης. Ε, και πόσο σημαντικό είναι και το στοιχείο τη πληροφόρηση προ του καταναλωτέ για να κάνουν εμπεριστατωμένα και έχοντα πλήρη επίγνωση κατάσταση την επιλογή του, Θα υποβάλω και εγώ κάποιε τροπολογίε για να συμπεριληφθούν στην ήδη άρτια γνωμοδότηση της ε, Μαρίας Γκραπίνη και ελπίζω ότι επιτέλου η Ευρώπη θα εγγύψει ευρυθώ ε, σε έναν από του πιο σημαντικού κλάδου τη Ευρωπαϊκή οικονομία. Η κυρία Κέπχαρτ έχει τώρα Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για την πολύ καλή, ε, το πολύ καλό σχέδιο αυτό και νομίζω ότι όντω στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε, αν κοιτάξουμε γύρω μας, ε, είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, έχουμε μια, ένα μεγάλο πλούτο ε, πολιτισμών, τοπίων που θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν πιο γνωστά σε όλο τον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει πολύ τον ε, τουρισμό. Θα πρέπει σίγουρα λοιπόν να το πράξουμε αυτό. Και εδώ νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τους τομείς ε, τους οποίους και εσύ ανέφερες. Η ποιότητα της προσφοράς και η αξιοπιστία ασφαλώς. Η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες σε αυτό το οποίο προσδοκούν. Καλό λοιπόν είναι να σημειωθεί πρώτα στον τομέα αυτό. Είναι επίσης ε, ουσιώδες να υπάρχει αξιοπιστία τους ε, τομείς, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος πριν από λίγο, των ε, νέων προσφορών, των νέων πλατφόρμων στο διαδίκτυο, να είναι εγγυημένη η ποιότητα. Στη Γερμανία πριν από κάποιο καιρό, στη Βαβαρία, ξέσπασε μία πυρκαγιά σε ένα σπίτι όπου φιλοξενούνταν τουρίστες και εκ των υστέρων προέκυψε ότι δεν υπήρχε άδεια για υποδοχή τουριστών, αλλά, εν πάση περιπτώσει, έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι πολίτες, οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι τουρίστες να είναι αξιόπιστες. Να ξέρουν ότι μπορούν να στηρίζονται σε αυτά που διαβάζουν, μεταξύ άλλων και για θέματα ασφαλείας ασφαλώς. Θα πρέπει λοιπόν να, συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε για διάφορα στοιχεία, να λάβουμε αποφάσει. Τρίτο και τελευταίο σημείο το οποίο ήθελα να αναφέρω και η ασφάλεια των εργαζομένων στους κλάδους αυτούς. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί ασφαλώς η ποιότητα παροχής υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς αντιμετωπίζεται ο υπάλληλος που παρέχει την υπηρεσία. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γκέπχαρτ και τώρα να δώσω το λόγο στον Άνταμ Ζάινφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επί, επί τη ευκαιρία να συμφωνήσω με τους ε, πολλούς συναδέλφους που είπαν ότι δεν αναγνωρίζεται δεόντως ε, ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτιμάται κάπως η αξία του και κακός. Αλλά ισχύει αυτό και μάλιστα έχει πολλά αίτια αυτή η υποτίμηση του τουρισμού. Ο κοινό πάντως παρανομαστής αυτής της ε, υποτίμησης είναι η, η περιθωριακή θέση που μερικές φορές δυστυχώς δίνουμε στον τουρισμό. Επίσης ε, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη το γεγονός ε, της Επιτροπής Μεταφορών που είναι καθήλη αρμόδια για το θέμα αυτό. Κάτι που είναι ενδεικτικό του, της υποτίμησης που διχάνει ο τουρισμός, γιατί οι μεταφορές είναι υποδομή. Ποια είναι το επίκεντρο του τουρισμού? Το ξενοδοχείο, που είναι το βασικό στοιχείο της ε, τουριστικής επιχείρησης. Οι υποδομές, οι μεταφορές ε, δεν είναι το θεμέλιο ε, του τουριστικού κλάδου, αλλά ένα τεχνικό στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το χαρακτήρα της υπήρου μας, τις πολιτιστικές μας αξίες, τις ιστορικές μας παραδόσεις. Ο τουρισμός είναι ένας βιομηχανικός κλάδος. Υπάρχει μια τουριστική βιομηχανία. Δεν είναι μόνο θέμα αναψυχής έχουμε και το θέμα το επιχειρηματικό, το βιομηχανικό. Και μερικές φορές, ε, ακόμη και οι πολιτικοί, ε, αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως ανάπαυλα, ως αναψυχή, ως διασκέδαση. Ε, δεν σταματάει ο τουρισμός στις διακοπές. Είναι σημαντικός τουριστικός κλάδος. Είναι πραγματική, πραγματική βιομηχανία. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο υπό τη σκοπιά της αναψυχής. Είναι πολύ σημαντικός κλάδος της οικονομίας. Είναι κρίμα να υποτιμάται. Κάτι που συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε ε, να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι έχει πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ο τουρισμός ε, και θα έχει ακόμη μεγαλύτερη αν τον αντιμετωπίζαμε σοβαρά και του δίναμε την αξία που έχει ως ε, τουριστική δηλαδή, ως βιομηχανική, βιομηχανικό κλάδο και όχι μόνο ως κλάδο της αναψυχής. δεν έχουμε μόνο ε, το, τον τουρισμό για λόγους αναψυχής, μερικές φορές γίνεται για λόγους που σχετίζονται με τον αθλητισμό και ούτω καθεξής. Οπότε θα πρέπει να φτάσουμε στον πυρήνα αυτού του κλάδου. Ε, δυστυχώς μέχρι στιγμής πολύ επιφανειακά ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Μόνο με την επιφάνεια. Και το αποφεύγουμε. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε επί τη ευκαιρία τα βασικά προβλήματα του τουρισμού που δεν επισημαίνονται δεόντως. Ένα άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι η προστασία των καταναλωτών, αλλά και το θέμα το τουριστικό και το οικονομικό. Και από αυτή την άποψη, ακριβώς επειδή ο καταναλωτής είναι στο επίκεντρο του κλάδου αυτού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δική του θέση και τα δικά του δικαιώματα. <coughs> Ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα ω Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ω μεμονωμένα κρατημέλη να έχουμε μια κοινή πολιτική για την προστασία και τη διάσωση μερικέ φορές των τουριστών και των καταναλωτών. Γιατί πολλέ φορές ε, οι τουρίστε ε, είναι εκτεθειμένοι στι επιθέσει, στην τρομοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και ίσως θα πρέπει να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να τα ρυθμίσουν. Επίσης, ε, γύρω από τον τουρισμό περιστρέφονται πολλά ε, επαγγέλματα που είναι ρυθμισμένα επαγγέλματα, κλειστά. Επίσης, ε, στην, η Πολωνία είναι κατηγορούν πρωταγωνιστή στο θέμα της απορρίθμισης των επαγγελμάτων. Αλλά δεν το κάνουν αυτό όλες οι χώρες. Σε πολλές χώρες έχουμε ρυθμισμένα επαγγέλματα και παθολογικότητα σε ό,τι αφορά την τα ρυθμισμένα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό. Κάτι τέτοιο είναι επιζήμιο και για τους επιχειρηματίες και για τους ίδιους καταναλωτές. Αυτή η υπερβολική ρύθμιση των επαγγελμάτων για τον τουρισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σανθόλ. Να πω δύο λόγια κι εγώ. Καταρχάς συμφωνώ ο τουρισμός πρέπει να θεωρείται ότι είναι πυλώνας της οικονομίας μας και όχι μόνο αναψυχή. Κάτι άλλο πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προσθέσουμε αξία και τι μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Και θεωρώ ότι αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, το ζήτημα της ασφάλειας και του ε, κατάλληλου ελέγχου να ε, εφαρμόζονται οι κανόνες. Ε, αλλά αυτό είναι από στα κράτη-μέλη, πιστεύω. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την προστασία των τουριστών ε, σε τρίτες χώρες. Ε, στην προηγούμενη θητεία κάναμε μια έκθεση για αυτό, για την επέκταση της ε, προξενικής προστασίας για Ευρωπαίους πολίτες και για πολίτες άλλων κρατών σε μια τρίτη χώρα, αλλά το Συμβούλιο το είδε εντελώς αρνητικά ενώ το Κοινοβούλιο το είχε δει θετικά. Ήδη κάποια κράτη-μέλη το κάνουν από μόνα τους, όπως οι βόρειες χώρες ναι, αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ιζαμπέλα Ντελμόντε που είναι ουσιαστικά η συγγήτρια της ε, έκθεσης αυτής ε, στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την συγγήτρια και όσου συμμετείχαν ε, στι εργασίε και στις συζητήσει από αυτή την Επιτροπή. Η συζήτηση αυτή αφορά ένα σημαντικό ζήτημα, το έχουμε υπογραμμίσει πολλέ φορέ. Ε, αναφερόμαστε σε μια τρίτη ευρωπαϊκή οικονομία, αναφερόμενη στον τουρισμό. Ποτέ δεν λέμε αρκετά για τον τουρισμό. Πρόκειται για ένα τομέα ευρύτατο στην ακρόαση που κάναμε. Μάθαμε ότι υπάρχουν 140 τύποι τουρισμού. Είναι ένα, υπάρχουν δηλαδή τύποι τουρισμού που ανήκουν σε, που απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ε, ομόν. Γίνεται λοιπόν όλο και πιο ιδιαίτερο ο τομέας αυτός και εξελίσσεται ραγδαία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την εισηγήτρια για τις προτάσεις, για την γνωμοδότηση και για τα όσα υπογράμμισε όσον αφορά τις θεωρήσεις, ε, τα διάφορα προσόντα ε, και, συγγνώμη, και, τα διάφορα, και τις διάφορες ενεργειακές πτυχές για να έχουμε έναν ε, βιώσιμο τουρισμό υπεύθυνο περιβαλλοντικά. Αναφέρθηκε επίσης και στα θέματα ποιότητας και αξιοπιστίας ε, για το οποίο έχει εκφράσει ήδη ε, άποψη η Ευρώπη στο πλαίσιο των τουριστικών επιχειρήσεων. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ναι, σίγουρα μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, αυτόν τον τομέα, ο οποίος ανθίσταται και στην κρίση. Προσφέρει θέσεις εργασίας σε γυναίκες, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε νέους. Ολοκληρώνοντας, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο sharing economy ε, που έχει συζητηθεί πολύ τελευταία. Ε, έχει δημιουργηθεί αυτή η έννοια της αρετής αυτής το sharing economy θα πρέπει να προστατευτεί εφόσον υποστηρίζει αυτή την αρετή, την κοινή χρήση, τον καταμερισμό μόλις γίνει κάποια δραστηριότητα παράλληλη με την επαγγελματική θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην νομοθεσία μαζί με τις επαγγελματικές δραστηριότητες. Συμφωνώ με τα όσα ακούσαμε προηγουμένως. Σίγουρα δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις καινοτομίες αλλά πρέπει να ρυθμίζεται και ο επαγγελματισμός και θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητε ε, διασφαλίσεις ε, όπω και για τι παραδοσιακέ δραστηριότητε. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά ειλικρινά να εκφράσω τι ευχαριστίε μου και πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να επανεκκινηθεί η σπουδαιότητα του τουρισμού. Είμαστε μεν ο πρώτος ε, παγκόσμιος προορισμός αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα ό,τι μπορούμε ώστε αυτή η ευκαιρία που έχουμε σήμερα να παραμείνει στο μέλλον όπου θα συνεχίσει να αυξάνεται σε απόλυτου αριθμού ο αριθμό των τουριστών. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε επαγγελματισμό και να εργαστούμε εντατικά ώστε ο τουρισμό να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ την ε, συνεισηγητρία από την Επιτροπή Μεταφορών. Δεν ξέρω αν η κυρία Ραπενή θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συζητητές και τους συναδέλφους που πήραν ε, το λόγο. Χαίρομαι που το σχέδιο έκθεση αυτό συγκέντρωσε τόσο μεγάλη προσοχή. Και ελπίζω να υπάρξει μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους κοιότητες εισηγητές σύντομα μετά την εξέταση των τροπολογιών και είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε να πετύχουμε συμβιβασμό προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κρατηθεί. Όλα όσα ακούσαμε εδώ σήμερα είναι σωστά και ορθά και θα πρέπει να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε μέσα στον τρόπο προκειμένου να μπουν στι τροπολογίε. Δεν είναι πολιτικό το παιχνίδι, να πούμε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να το κοιτάμε από οπτική γωνία πολιτική ομάδα. Όχι. Αυτό που μα ενώνει είναι το συμφέρον του κλάδου σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να αναζητήσουμε νέε μεθόδου, νέα εργαλεία για νέα ανάπτυξη στον τουρισμό. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το θέμα δεν είναι μόνο οι διακοπές. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και την, τον πολιτισμό, την επαφή με τον πολιτισμό άλλων και στη Ρουμανία όταν ήμουν υπουργό πολιτισμού πρέπει να σας πω ότι έμαθα πολλά καινούργια πράγματα για την ίδια τη χώρα. Πολλά λοιπόν μπορούν να μάθουν οι πολιτέ για την χώρα τους, πόσο μάλλον και για τις άλλες χώρες της Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για χώρες με πολύ πλούσιο τουριστικό δυναμικό και είμαι πεπισμένη ότι η έκθεση, η γνωμοδότηση τελικά θα μας ε, βρει όλους σύμφωνος. Χαίρομαι λοιπόν για την έκθεση αυτή και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τονίσουμε όλες τις πτυχές ε, των σκιατών εισηγητών από πλευρά της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Δεν είμαστε από την Επιτροπή ε, μεταφορών, εμάς μας απασχολούν τα στοιχεία που άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη την ποιότητα των ε, εργασιακών εθνικών των υπηρεσιών που παρέχονται, την εμπιστοσύνη στον ε, τουρισμό στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους σας και είμαι βέβαιη ότι θα συνεργαστούμε εξαιρετικά με τους κοιότητες εισηγητές για να είναι τελικά καλή έκθεση και να ληφθούν υπόψη οι απόψει όλων όσοι πήραν το λόγο σήμερα. Και το έγγραφο αυτό ελπίζουμε ότι θα μα βοηθήσει στο μέλλον. Γιατί αν δεν έχει κάποια πρακτική εφαρμογή το έγγραφο αυτό, δεν έχει νόημα. Να σα πω επίση ότι επειδή είμαι τον ιδιωτικό κλάδο πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ λέει η πρόεδρο. Ελπίζω να μα βοηθήσει όλου να αντιμετωπίσουμε τον τουρισμό με την αξιοπρέπεια και με τη σημασία που του αρμόζει στην πολιτική συζήτηση. Χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τροπολογίε 24 Ιουνίου στι 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση αυτή για τον τουρισμό και τώρα θα περάσουμε στην νομοδότηση για την μείωση των εκπομπών ρήπων από οδικά οχήματα. Η Ρούσα Τουν Χόλτμαν είναι η εισηγήτρια. Ο Άλμπερ είναι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, ο εισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω από 60 τροπολογίες έλαβα για την γνωμοτοδοσία αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες αυτές τις τροπολογίες. Για κάποιες από αυτές μπορώ να σας πω ότι με χαρά μου θα τις υποστηρίξω. Για κάποιες άλλες ωστόσο θα ήθελα να τις συζητήσουμε. Συγκεκριμένα. Να αναφέρω ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες πάνω από 20 στην αριθμό που διαγράφουν την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να κάνουμε τέτοιες ανακλήσεις. Δεν πληροφορήθηκα στις εργασίες μου προετοιμασίας του εγγράφου και στις συζητήσεις μου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επρόκειτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεκτείνει την ε, εντολή της. Ένα μόνο ζήτημα υπάρχει, όπου στην πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά επιπλέον εξουσίες αμμοδιότητες για το διοξίδιο του αζότου σε ό,τι αφορά και τις ε, κρύες θερμοκρασίες. Τις δοκιμές σε ψυχρές ε, θερμοκρασίες. Κάναμε λάθος γιατί υποτιμήσαμε τις συνέπειες ε, του εκπομπών διοξιδίου του αζότου στην ε, ατμοσφαιρική ποιότητα και στην υγεία μας. Θα πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε αυτό, γιατί η ρήπανση και οι συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου είναι πραγματικά δραματικές σε κάποιες περιπτώσεις και θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερα στοιχεία εδώ πέρα. Κατά δεύτερον, να πω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ τεχνική φύσεω και πραγματικά δεν θα πρέπει να δώσουμε πολιτική διάσταση. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω να δώσουμε ε, εντολή και αρμοδιότητα στην Επιτροπή προκειμένου να μπορεί να δράσει και θα ήμουν κατά τη διαγραφή κατά των τροπολογιών που προτείνουν διαγραφή. Δύο τροπολογίε τώρα ήταν να μην συμπεριληφθεί το μεθάνιο στις ε, εκπομπέ αυτέ διεξοδία του άνθρακα. Είμαι ανοιχτή σε συζητήσει. Υπάρχει η πρόταση των σοσιαλιστών και δημοκρατών για την κατανάλωση μετρητές κατανάλωσης καυσίμων. Εγώ είχα κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά η διαφορά είναι ότι εγώ είχα προτείνει να γίνουν αλλαγές σε ό,τι αφορά τους μετρητές κατανάλωση καυσίμων τώρα και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις για τους δείκτες αλλαγής ταχύτητας. Σε ό,τι αφορά τις ε, τις δείκτες, ε, τις μετρητές ε, κατανάλωσης ε, καυσίμων, μπορούμε να το περάσουμε τώρα. Αν συμφωνείτε λοιπόν, μπορώ να προετοιμάσω σχετικέ τροπολογίε. Κάποιε άλλε τροπολογίε είναι υπερβολικά τεχνική φύση ή επισέρχονται σε τομεί που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα γίνει συνάντηση των σκιονδών στι 9 Ιουνίου. Και στην περίσταση αυτή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε εκ νέου τι τροπολογίε. Στη συνέχεια στις 22 και 29 Ιουνίου. Αυτά λοιπόν είχα να αναφέρω α, για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε την εισηγήτρια και τώρα να δώσουμε το λόγο στους κοιότης από πλευρά της Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Πολύ χρήσιμες οι σκέψεις σας ε, για πολλές ε, από τις τροπολογίες και τα θέματα που επισημαίνουν. Είμαστε υπέρ των μέτρων που συμβάλλουν στη μείωση των ρήπων των εκπομπών ε, αερίων και τη βελτίωση της ε, ποιότητας του αέρα. Συμφωνούμε απόλυτα λοιπόν. Και είναι σημαντικός αυτός ο κίνδυνος ε, της ατμοσφαιρικής ρήπανσης για την ανθρώπινη υγεία. Και υπάρχουν όλο και περισσότερα τεκμήρια για αύξηση των κινδύνων. Και παρόλο που βελτιώνουμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε επιζήμια ακόμη αποτελέσματα στην υγεία και στο Λονδίνο, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Πολύ συχνά έχουμε υπέρβαση των ορίων των οξυδίων του, του αζότου και του διοξιδίου του αζότου. Έχουμε ξεπεράσει τις οριακές τιμές ήδη τη δεύτερη μέρα του χρόνου στο Λονδίνο. Και είμαστε υπέρ των ευρωπαϊκών δράσεων για να καθοριστούν περαιτέρω αποδεκτές ε, ε, οριακές τιμές για τις τοξικές ε, ουσίες, τα τοξικά αέρια και τα καυσαέρια και την καλύτερη ευθυγράμμιση της κοινοτικής νομοθεσίας. Αντιλαμβάνομαι ε, τις ε, επιφυλάξεις και τις ανησυχίες μας ό,τι αφορά την πρόταση για τις κατεξοδότηση πράξεις. Εμείς προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τη διατύπωση που περιλαμβάνεται και το, τις διατάξεις για τις κατεξοδότηση πράξεις. Την παράταση με, με την αύξηση ή την ε, ανάκληση σε ό,τι αφορά τις και τι σχετικέ αρμοδιότητε. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πάντω λύση και να συνεννοηθούμε για το θέμα των κατεξουδότηση πράξεων. Θεωρώ ότι έγινε σημαντική πρόοδο ε, για το περιεχόμενο τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή ΣΥΜΚΟ και θα θέλαμε ε, να δούμε τη κανονική χρήση, γιατί πολλές δοκιμές γίνονται με βάση την κανονική χρήση των οχημάτων και χαίρομαι που σχολιάσατε τις ε, προτάσεις μας για τις ενδείξεις ε, αλλαγές ταχύτητας και την ανάγκη να, τα, να τους ε, συμπεριλάβουμε σε αυτά τα μέτρα. Επίσης, έχουμε σοβαρές ανησυχίες ε, για την έκθεση της ΕΜΒΗ, που είναι η αρμόδια ουσίαν επιτροπή. Και έχουμε στενή συνεργασία ε, με τους σκιώδες και τον υπόλοιπων και των άλλων ε, δύο επιτροπών, ΕΜΒΙ και ΤΡΑΝ, ώστε να επηρεάσουμε θετικά την κύρια έκθεση. Γνωρίζω ότι είναι τεχνική φύσεως η έκθεση, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντική. Και τέλος θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και μάλιστα κάπως πιο διεξοδικά το θέμα του μεθανίου. Ευχαριστώ κύριε Άντερσον από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές, ο κύριος Ντάλτον. Ευχαριστώ πολύ για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ε, καλωσορίζω πολλά τα στοιχεία εδώ. Θα διευκολυνθούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων από νομοθετική άποψη, θα τους δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία. Ειδικότερα αναφέρεσουμε αφαιρέσουμε τις δύο διαφορετικές εγκρίσεις τύπου, είναι καλή κίνηση. Η πρόταση επίσης ε, απορρίψης ε, των ορίων αμμονίας για τα βαρέα οχήματα είναι καλή. συμφωνώ με την Κομισιόν για τις ε, εκπομπές διοξιδίου του αζότου, αλλά βασικό από την ομάδα μας στο σχόλιο, θα το δείτε από τις πολλές τοπολογίε που έχουν υποβάλει τα μέλη του UCR, e είναι το ζήτημα των κατεξοδότηση και εκτελεστικών πράξεων σε σχέση με τη βασική πράξη. Η δική μας άψη γενικά είναι ότι από παρελθούσα εμπειρία στην προηγούμενη θητεία μάθαμε ότι αν θέλουμε πραγματικά το κοινοβούλιο να ε, παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε τέτοια νομοθετήματα πρέπει να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στη βασική πράξη. Η εκχώρηση αυτή εξουσιών αποδυναμώνει το Κοινοβούλιο και τους συνομοθέτες. Καταλαβαίνω φυσικά όταν είναι τεχνικά τα ζητήματα, αλλά ορισμένα από αυτά τα ζητήματα είναι εξίσου πολιτικά. Ε, το να επαναταξινομήσουμε το μεθάνιο ως ε, ε, εκπομπή ε, ως αέριο του θερμοκηπίου θα πρέπει να υπάρχει στη βασική πράξη. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε σε τη εκτελεστική πράξη το ίδιο για τις εκπομπές διοξιδίου του αζότου. Πρέπει να συζητάμε, πιστεύω, ποιο θα είναι το όριο ε, μέσω συναπόφασης και πρέπει να συμπεριληφθεί στη βασική πράξη. Ε, θεωρώ ότι αυτή γενικά, γενικά την πορεία πρέπει να ακολουθούμε εγώ είχα διαπραγματευτεί την μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική την προηγούμενη θητεία και ένα μήνα περίπου αφού ολοκληρώσαμε τι διαπραγματεύσει, καταλάβαμε πόσα χάσαμε όταν η Κομισιόν άρχισε να προβάλλει διάφορε εκτελεστικέ και κατεξουδότητε πράξει και εκεί καταλάβαμε και, για τι οποίε εμεί δεν έχουμε και πολλά να κάνουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε πραγματικοί συνομοθέτες και να αναγνωριζόμαστε ω τέτοιοι, θα πρέπει να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στη βασική πράξη, παρότι κάποια από αυτά τα ζητήματα είναι αρκετά τεχνικά. Έχουμε πιστεύω την εμπρογνωμοσύνη για να το πράξουμε. Ευχαριστώ κύριε Ντάλτον. Δίνω το λόγο στην κύριο Ροσφόρ για την ομάδα Άλντε. Ευχαριστώ κύριε... Πρόεδρε, η σκιωδή συγγήτρια ήταν εδώ στην ψηφοφορία, αλλά έχει φύγει, διότι μας εκπροσωπεί στην ε, συνέλευση με την, Ευρωπαϊκή, με την Λατινική Αμερική. Ε, Ανέφερε λοιπόν να σας μεταδώσω το μήνυμά της που σχετίζεται με τη συζήτηση που κάνουμε εδώ και μερικά λεπτά. Σας το διαβάζω. Καλωσορίζουμε τη δέσμευση όλων των μερών για περαιτέρω μείωση των εκπομπών οδικών οχημάτων. Αποτελεί μια πρόκληση που όλοι δεχόμαστε. Αυτό που δεν μπορεί να δεχθεί η συνεισηγητρία είναι η νομική μορφή που ζητείται από αυτή την πρόταση. Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ε, ανθίστατος ορισμένες προσπάθειες ε, απόσυρσης εξουσίας από το Κοινοβούλιο ε, προς όφελος της Κομισιόν μέσω κατεξιοδότηση και ε, εκτελεστικών πράξεων. αυτό αφορά δύο ανοιχτού διαλόγου τουλάχιστον. Δεν καταλαβαίνει γιατί η Επιτροπή μα να υποστηρίξει κάτι τέτοιο εδώ, ενώ αντιτίθεται σε αυτό σε άλλα θέματα, σε άλλε γνωμοδοτήσει. Γι' αυτό το λόγο υπέβαλε τόσε πολλέ ε, ε, τροπολογίε διαγραφή του κειμένου. Σύμφωνα με του γλωσσομαθεί νομικού, δεν υπήρχε δυνατότητα να αλλάξουμε το Delegation Act σε Ordinary Legislative Procedures σε τόσες πολλές περιστάσεις. Αντί γι' αυτό η Κομισιόν θα πρέπει ήδη να προσθέσει τις δικές της τεχνικές ε, ε, τροποποίησεις, τροπολογίες στο κείμενο και καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν η συνεισηγητρία θα ζητήσει από την Κομισιόν να επανεπεξεργαστεί την πρόταση και να την ξαναεποβάλει όταν θα είναι έτοιμη με όλες τις τροπολογίες με τα όρια εκπομπών στη νέα πρόταση. Κάνοντας αυτό είναι πολύ πιθανό να, η συνεισηγητρία να αντιδραστεί διαφορετικά στο κείμενο. Ευχαριστούμε κύριε Ροσφόρ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέρφους αν επιθυμούν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Δεν βλέπω κανέναν, οπότε ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ανοίξετε και το μικρόφωνο σας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους, συνα... τους ευρωβουλευτές για τις τροπολογίες που κατέθεσαν και την εισηγήτρια. Πρώτα απ' όλα, και να υποβάλω κάποια σύντομα σχόλια για την εκχώρηση εξουσιών, για τις κατεξοδότηση πράξεις. Σας διαβεβαιώ ότι πρόκειται για τεχνικά θέματα μόνο. Και το πρόβλημα που βλέπουμε στην ατμοσφαιρική ρήπανση στην Ευρώπη είναι οξύ. Η ποιότητα του αέρα είναι μείζον ζήτημα και χρήζει άμεσα αντίδρασης, ταχείας αντίδρασης από πλευράς νομοθετών. Οπότε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να, να υποβάλει πρόταση ε, με την κανονική διαδικασία και τα συνοδευτικά έγγραφα, η διαδικασία αυτή θα είναι χρονοβόρα, οπότε θα εξουδετερωθεί η ανάγκη της ταχείας αντίδρασης για τη βελτίωση της ατμοσφαιρικής ρήπασης. Γι' αυτό ζητήσαμε κατά εξουσιοδότηση πράξης. Οπότε για αυτές τις πράξεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, παρόλα αυτά θα έχει σημαντική επιρροή στην τελική μορφή της πρότασης. Στη θέση σας ε, δεν θα ανησυχούσα για περιορισμό των ε, αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε περίπτωση που υιοθετηθεί αμετάβλητη η πρόταση του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρούζα, θα ήθελες να δευτερολογείς για να ολοκληρώσουμε. Δύο λόγια μόνο γιατί θα έχουμε πολλές ευκαιρίες. Θα συναντηθούμε σε 9, στις 22, στις 29 Ιουνίου. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να ξανασυζητήσουμε. Τώρα, η εξοδότηση αυτή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημαίνει ότι αποποιούμαστε την επιρροή μας αλλά είναι θέμα ζωής και θανάτου γι' αυτό και ο χρόνος είναι πολύτιμος και η ταχεία αντίδραση είναι επιτακτική ανάγκη και συμφωνώ με την έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση αυτών, αυτής εξουσιοδότησης. Ευχαριστώ τους ε, σκιώδης ηγητές για την ε, καρποφόρα συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί και με αυτήν ήταν επικοδομητική συνεργασία. Ε, ευχαριστώ τον Λούκα Σενόφσκι, τον Βίκτορ που επέστρεψε στη γραμματεία και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Και ας μην ξεχνούμε συνάδελφοι αυτό το θέμα των ρήπων αλλά κυρίως των ρήπων υπό το πρίσμα της υγείας, γιατί έχουμε πραγματικά εντυπωσιακά νέα επιστημονικά πορίσματα και έρευνες για το θέμα αυτό. Θα συνεχίσουμε τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών στις 22 και 23 Ιουνίου, ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ στις 29 Ιουνίου. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση επί της γραμματότητας για τη μείωση των ρήπων από τα οχήματα. Περνάμε τώρα στην έκθεση σε ό,τι αφορά την καλύτερη ρυθμίση της ε, ενιαίας ε, αγοράς. Η, η Ανελή είναι η συγκεκριά μας. Έχει το λόγο, Ανελή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τον Απρίλιο, ε, τον Απρίλιο σας παρουσίασα το σχέδιο έκθεσης για την καλύτερη νομοθεσία και χαίρομαι λοιπόν που σήμερα ε, μπορώ να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης, το επίσημο πλέον. Να ευχαριστήσω τους κοιόδους συζήτητες οι οποίοι έκαναν τις πρώτες παρατηρήσεις τους ε, στο σχέδιο εργασίας, το γράφο εργασίας και θα τις λάβουμε υπόψη. Και εγώ θα ήθελα να σας πω την αλήθεια να έμπαιναν πιο πολλά στοιχεία στο κείμενο, αλλά δεν είχαμε και δυνατότητα να επεκτείνουμε το κείμενο. Το σχέδιο έκθεσης έχει ως βασικό στόχο να υπάρχει καλή, απλή, διαφανής νομοθεσία για να εγγυηθεί την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη που να δώσει όθεση με τη σειρά τη ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό είναι ο απότερο στόχο. Μια Ευρώπη η οποία δεν απογοητεύει, αλλά η οποία δίνει κίνητρα. Και ξεκινάμε λοιπόν με βασική αρχή την επικουρικότητα. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σημαντικό καθήκον και για τα τρία θεσμικά όργανα, για το Κοινοβούλιο, αλλά και για την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και για τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τα οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή και έχω ιδιαίτερο υπόψη μου το γεγονό ότι δεν έχουν ουσιαστικά χρόνο για να κρίνουν την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, τήρηση ή μη τη αρχή ε, τη επικουρικότητα. Προτείνω λοιπόν να του δώσουμε πιο πολύ χρόνο. Επίση, ε, με τη διαδικασία κόκκινη κάρτα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που δεν τηρείται η αρχή της επικούρικότητα Στο σχέδιο έκθεσης επίσης αναφέρονται και κάποια συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία προτείνονται, για να πετύχουμε την καλύτερη νομοθεσία. Καταρχάς η μελέτη αντικτύπου Impact Assessment πολύ έχει συζητηθεί και ο Φραν Τίμερμαν το συζητάει και το έχει παρουσιάσει στην ε, παρεμβάσεις του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι μελέτες αντικτύπου να θεωρούνται έγγραφα ζωντανά που εξελίσσονται. Φυσικά θα πρέπει να προσαρμόζονται στις μεγάλες αλλαγές, να μην υπάρχει γραφειοκρατικό άχθος, να βασίζονται σε επιστημονικά τεκμήρια και επιστημονικές γραμματοτήσεις, evidence-based και επίσης για την ε, αξιολόγηση των ε, μελετών αντικτύπου θα πρέπει το Scrutiny Board που θα αποτελείται από Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο να συμπεριλαμβάνει και κάποιους α, ε, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Επίσης, η, το σχέδιο έκθεσης ε, προτείνει καλύτερη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να δώσουμε σε όσο πιο πολλούς γίνεται τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους. Να μην είναι μεγάλα εμπόδια για τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων. Ένα φόρουμ εμπλεκομένων φορέων θα ήταν μια αρμόζουσα λύση, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά. Επίσης, τίθεται θέμα της εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων και η καλή εφαρμογή σε διάφορα κράτη-μέλη σήμερα είναι ένα πρόβλημα. Και το Βέλγιο σίγουρα είναι και συγκαταλέγεται στους κακούς μαθητές. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από το... την πατρίδα μας πάντα. Είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακολουθεί την εφαρμογή και να επιλύει τα προβλήματα από αυτά ανακύπτουν. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, πρέπει να κάνει πιο πολλές προσπάθειες σε ό,τι αφορά Ενδεχομένω ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον έγκαιρο εντοπισμό προβληματικών τομέων για τα κράτη-μέλη στην επόμενη φάση, τα οποία δεν ε, εφαρμόζουν την νομοθεσία, θα πρέπει να υπάρχει πιο συστηματική αντιμετώπιση. Και εδώ πρέπει να δώσουμε πιο πολύ προσοχή στις ε, παραβιάσεις εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο. Τέλος, το σχέδιο έκθεσης ε, αναφέρεται και στην σημαντική τελική φάση της νομοθεσίας, την αξιολόγηση και την ενδεχόμενη αναθεώρηση των κανόνων. Διαρκώς λοιπόν θα πρέπει να κοιτάμε κατά πόσον οι φυσάμενοι κανόνες εκπληρώνουν τον στόχο για τον οποίο καταρτίστηκαν. Κατά πόσον εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι. Γιατί συχνά ακούμε ότι η συσσόρευση του κόστους όλων των κανόνων δημιουργεί τελικά προβλήματα για τις μικρές επιχειρήσεις και για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αυτά ήταν συντομία τα πιο σημαντικά στοιχεία στο σχέδιο έκθεσης. Πιο πολλές λεπτομέρειες ασφαλώς θα βρείτε στο ίδιο το κείμενο και προσβλέπω στις ε, τροπολογίες που θα λάβω. Δεν είμαι σίγουρη για το χρονοδιάγραμμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μας βοηθήσει η γραμματεία σε ό,τι αφορά την προθεσμία, δηλαδή. Δέκα, 9, εννέα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια. 9 Ιουνίου είναι η προθεσμία, πράγματι, και τώρα θα αλλάξουν και θα γίνω συνεισηγήτρια για το ΕΛΚ. Θα μιλήσω ω συνεισηγήτρια του ΕΛΚ. Καλώς ορίζω την έκθεσή σας. Αληθεύει ότι έχουμε καταμερισμένη ευθύνη για βελτιωμένους κανονισμούς ώστε να προσφέρουμε περισσότερη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρε ο Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμαντς ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μεγάλο τρόπο τα μεγάλα πράγματα και μικρό τα μικρά δεν αφορά τη μείωση των δικαιωμάτων αλλά της γραφειοκρατίας το όλο θέμα. Μείωση της γραφειοκρατίας. Εξάλληψή της. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να δούμε πώς ε, η νομοθεσία μας ε, θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και η νομοθεσία μας βέβαια είναι πάντα συμβιβασμός. Ο συμβιβασμός μας πολλές φορές είναι τόσο ακατανόητος, δυσνόητος, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες. Αυτός λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, πρέπει να είναι ο στόχος μας. Κάπου χάσαμε την έκθεση ΣΦΑΜΠ για την ε, διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και τη γνωμοδότηση της ΣΥΜΚΟ ως παραπομπή. Και τώρα επί της ουσίας ε, εγώ είμαι επιφυλακτική για τις κόκκινες κάρτες. Δεν πιστεύω ότι τα κοινοβούλια πρέπει να υποβάλουν βέτο το ένα στο άλλο. Πρέπει να έχουμε, ε, να συνδιαλεγόμαστε. Όπω μα επιτρέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα, και δεν το έχουν καταλάβει πολλοί, η συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει περισσότερε εξουσίε στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, στο πλαίσιο της νομοθετικής μας διαδικασίας. Όπως έχουμε λοιπόν σε διάφορες άλλες εκθέσεις, αυτό μπορούμε να το ενισχύσουμε, να έχουμε ε, εκ των προτέρων διάλογο, ειδικότερα για τις οδηγίες στα ε, εθνικά μας κοινοβούλια, να τα εμπλέκουμε περισσότερο και εδώ, πράγμα που ήδη προσπαθούμε να κάνουμε, αν και συχνά δεν παρίστανται για διάφορους λόγους, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Κατά την όψη μου, δεν είναι καθόλου επικοδημητικό να καταναλώνουν τον περισσότερο χώρο, τα, χρόνο τα, εθνικά κοινοβούλια σε δοκιμές επικουρικότητας. Πρέπει να συμμετέχουν απλά σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα για την εκτίμηση αντικτύπου είναι κάτι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η ψηφιακή επανάσταση, η ψηφιοποίηση και φυσικά η νομοθεσία μας θα πρέπει να προβλέπει πράγματα και για το μέλλον, για πράγματα που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Ξέρετε, η ψηφιακή επανάσταση κινείται ταχύτερα από την πολιτική. Δεν πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Διαρκώς μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και συμφωνώ ε, αλλά εκεί που λέτε ε, πρέπει να αλλάξουμε λίγο ξέρετε, την σύνταξη, ίσως να είναι γλωσσικό το θέμα εκεί που μιλάτε για την ανταγωνιστικότητα και τους πολίτες. Ε, και εκεί που λέτε living document, ε, ζωντανό έγγραφο, συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ζωντανό έγγραφο δεν σημαίνει μία ε, μεγάλη διαδικασία που παίρνει πολύ χρόνο, με πολλέ φάσει, με πολλά βήματα που το περιπλέκουν ακόμη περισσότερο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για βελτίωση της νομοθεσίας, μια νομοθετική διαδικασία πιο αποτελεσματική και όχι πιο περίπλοκη. Για το ζήτημα στην παράγραφο 10, το παράλληλο οργανισμό που θα μπορεί να σταματήσει να μπλοκάρει νομοθεσία, έχω σοβαρές επιφυλάξει αυτό. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να μειώσουμε να αποδυναμώσουμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που λειτουργούμε μεν, αλλά όχι να αφαιρέσουμε εξουσίες από όργανα υπεροργάνων που δεν έχουν νομική βάση ε, ύπαρξη όπως ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε τώρα όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή. Πολύ καλά τα λέτε. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και μια παραπομπή στα τα EU Sweeps ε, στην παρακολούθηση των ιστοσελίδων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό να παρακολουθούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη όντω ε, υλοποιούν ε, την υπάρχουσα νομοθεσία για την ψηφιακή αγορά. Και αυτό το Solving Plus, Plus το Solvit Plus πιστεύω είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον έλεγχο της εφαρμογής της ψηφιακής αγοράς και οι ψηφιακές πλατφόρμες όπως το ενημερωτικό σύστημα για την ψηφιακή αγορά και διάφορα άλλα. Όλα αυτά είναι συστήματα που επιτρέπουν την ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ κρατών μελών, την επιτάχυνση της υλοποίησης και επίσης έχουμε το EDR και το ODR ε, για την επίλυση διαφορών ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών και επίλυση διαφορών online. Έτσι αποφεύγεται ε, αποφεύγονται δικαστικές αγωγές είναι μια καλή λύση για πολίτες και για εταιρείε. Καλό θα ήταν να επιταχύνουμε την υλοποίηση. Τώρα, όσον αφορά τη μεταφορά, το πρόβλημα πιστεύω δεν είναι το πλήθο των μελετών. Το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε, μεταφέρεται η νομοθεσία, αλλά μετά πώ υλοποιείται. Και ξέρετε, η αξιολόγηση τη υλοποίηση είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο από την αξιολόγηση τη μεταφορά. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε δείκτες μέτρησης αξιολόγησης της υλοποίησης. Και ξέρετε, από αυτήν την άψη έχουμε τώρα το ευρωπαϊκό εξάμεινο και θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση για να αξιοποιηθεί ε, πλήρω, να συμπεριληφθεί η ενιαία αγορά, η ψηφιακή αγορά στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Έχω και άλλα ζητήματα που είναι λιγότερο σημαντικά τώρα. Θα μιλάτε για το κόστο και τα ωφέλη τη ενιαία αγορά ε, που θα γίνουν αισθητά από ποιον. Ε, έχετε κάποιες ενδιαφέρουσες σκέψεις για το σύστημα προώρης ειδοποίησης ε, να τα αναλύσετε λίγο παραπάνω δεν έχω κάποια διαφωνία τώρα όσον αφορά την επιβολή ξέρετε οι διαδικασίες κατά παραβάση ε, πρέπει να είναι ταχύτερες και να χρησιμοποιείται από την Κομισιόν χωρίς διπλά κριτήρια χωρίς άλλα μέτρα και άλλα στάθμα αναφέρεστε σε ενδιάμεσες διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να επιταχυνθεί από το δικαστήριο αυτή ε, ε, να, να, να, να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες κατά παραβάση, οι παίρνουν πολύ χρόνο. Τώρα για τις εξαγωγές, για τις εξαγωγές ε, θα πρέπει πιστεύω να βάλουμε τη δοκιμή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δοκιμή του ηλεκτρονικού εμπορίου στην έκθεση. Είναι δύο μέσα χρήσιμα που επιτρέπουν την αποφυγή του gold plating και των λάθος ερμηνεών. Όσον αφορά την ε, sunset clause και την υιοθέτησή της, συμφωνώ μαζί σας, είναι σημαντική αρχή, αλλά δεν μπορούμε να την έχουμε, να την αναφέρουμε αναφηρημένα. Πρέπει να σχετίζεται με κάτι πραγματικό, με κάτι που συμβαίνει πραγματικά, γιατί αλλιώς ε, θα, έχουμε τον, θα υπάρχει κίνδυνο να αφαιρέσουμε μια ρήτρα τέτοια τη Sunset Clause από την νομοθεσία χωρί να την αντικαταστήσουμε με κάτι. Οπότε ε, αναμένω να συνεργαστώ με εσάς και τους άλλους κοιόδης. Ε, είναι πολύ σημαντική πιστεύω αυτή η έκθεση, ειδικότερα αυτή την εποχή που η Κομισιόν δουλεύει για το ρηφίτ και τη βελτίωση της νομοθεσίας. Τώρα λοιπόν ξαναγίνομαι πρόεδρος και δίνω το λόγο στους, στους όδη ε, των σοσιαλιστών Κρίστο Σαλτεμόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, γιατί το σχέδιο γνωμοδότησή τη είναι πολύ καλύτερο στη σημερινή του μορφή. Και χαίρομαι που οι ενστάσει μας έλειψαν υπόψη. Έχω μερικέ γενικέ και κάποιες πιο ειδικέ παρατηρήσεις. Καταρχήν όλοι συμφωνούμε ότι η εσωτερική αγορά χρήζει καλύτερη νομοθεσία. Είναι προφανές. Αλλά εφνομοθετήν δεν σημαίνει αποφύγη νομοθεσία. Αν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα ότι το καλύτερο είναι η αδράνεια, ξεχάστε το. δεν θα πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχή της κόκκινης κάρτας, συμφωνώ εν μέρη με το σημείο 5, να παρατείνουμε τις προθεσμίες για, τη, για τις περιφερειακές και εθνικές βουλές, όχι μόνο για την κόκκινη, αλλά και για την κίτρινη κάρτα. Γιατί μερικές φορές είναι υπερβολικά σύντομες οι προθεσμίες για να εγγύψει κάποιος στην νομοθεσία. ξέρω τώρα θα πρέπει να τροποποιήσουμε τις θήκε για να μπορούμε να δίνουμε αυτόματα ε, κόκκινη κάρτα. Ίσως θα μπορούσαμε να παρατείνουμε τις προθεσμίες και να προβλέψουμε κίτρινη κάρτα. Τώρα, θα πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο των μέτρων. Αλλά μην ξεχνάμε και την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών. Σημείο 9. Πρόκειται για ένα έγγραφο δυναμικό, ζωντανό, όχι στατικό. Συμφωνώ επί της αρχής. Όπως είπα όμως και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, ένα ζωντανό έγγραφο δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια την ε, υπερβολική παράταση της νομοθετικής διαδικασίας. Γιατί ήδη είναι χρονοβόρα. Και αν ε, υπό το πρόσχημα της ε, ζωηρότητας και της ε, εξέλιξης, ενισχύσουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες, δεν πιστεύω ότι είναι αυτό ο στόχος. Και φυσικά και το έγγραφο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μακροσκελές. Σημείο 10. Ελεγκτικό όργανο. Έλεγχος των αναλύσεων και δυνατότητα ανάκλησης μιας απόφασης. Είμαι κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις συνέπειες των νομοθετικών μας μέτρων, αλλά αυτό να γίνεται από τους πολιτικούς. Μόνο αυτοί να μπορούν να ανακαλούν, να καταργούν νομοθετικές διατάξεις. Όχι ένας ανεξάρτητος ελεγκτικός ε, οργανισμός. Σημείο 11. Η διαδικασία ακρόασης των ενδιαφερομένων. Συμφωνώ, αρκεί να μην είναι υπερβολικά χρονοβόρη διαδικασία. Είναι σημαντικό οι stakeholders, οι ενδιαφερόμενοι, να γνωστοποιούν τις απόψεις τους αλλά να μην κρατάει στο δυναικές αυτή τη διαδικασία. Και γίνεται και μια πολιτική αξιολόγηση των συνεπειών και τον τελικό ρόλο λόγω να έχουν αντικειμενικά αντικειμενική και ανεξάρτητη εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ με τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά γιατί όχι να μην συμμετέχουν και οι πολίτες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, σημείο 18, το gold plating, αυτός ο κανονιστικός υπερθεματισμός. Συμφωνώ απόλυτα ότι όταν υποβάλλουμε ένα νομοθετικό μέτρο, μερικοί έχουν την τάση να υπερθεματίζουν και να προσθέτουν στρώματα. Θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο μόνο εφόσον είναι απαραίτητο. Γιατί μια οδηγία πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική ενωμή τάξη μερικές φορές χρειάζονται συμπληρωματικές διατάξεις για να ληφθούν υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες. Αυτό δεν σημαίνει κανονιστικό υπερθερματισμό, αλλά απλώ η λήψη υπόψη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Αυτά προς το παρόν. Επειδή υπάρχουν πολλά και διαφορετικά σημεία, θα μπορούσαμε να συζητούμε ώρες πολλές αλλά το βασικό είναι να φροντίσουμε να βελτιώσουμε την νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ωφελήσει και τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στον Λατούνες ε, που είναι σκιώδης από την Άλντε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ε, συνάδελφοι συγκήτρια. Πολύ καλή και πολύ επικοδομητική αυτή η έκθεση στο σχεδιό της. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχική συζήτηση τον Απρίλιο, συμφωνώ πολύ με τη γενικότερη γραμμή που ακολουθεί η έκθεση. Και πιστεύω ότι περιλαμβάνονται πολλά σημαντικά στοιχεία. Ιδιαίτερα η παράγραφη για την μελέτη αντικτύπου, για τη διαδικασία διαβούλευση και για την εφαρμογή γενικότερα. Πρόκειται για τομεί που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε τους, τον τρόπο λειτουργία τη νομοθεσία στον τομέα τη ενιαία αγορά. Μ' αρέσει επίση το γεγονό ότι τονίζεται την ενιαία αγορά ω παράγοντα δημιουργία θέσεων απασχόληση και ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί την πρώτη στην προτεραιότητα στην παρούσα φάση. Και επίση ε, με απασχολεί η ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν που αναφέρεται στο σχέδιο έκθεση. Είναι καλή λοιπόν η γνωμοδότηση, αλλά θα κάνω και κάποιες ε, προτάσεις βελτίωσης σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, θα ήθελα να οριστεί η ιδέα του φόρουμ των εμπλεκομένων φορέων, που αναφέρεται στην παράγραφο υπαρτιμών 14. Το ίδιο προτείνει και ο Επιτροπός Τίμερμαν σε ό,τι αφορά μια ένα φόρουμ ενδιαφερομένων μερών για το refit. Νομίζω ότι καλό θα είναι να αναπτύχθει λίγο παραπάνω ποιο θα είναι ο σκοπό του φόρουμ αυτό. Κάτι άλλο που ήθελα να προτείνω. Η, η ιδέα των σταθερών προθεσμιών εφαρμογής. Εδώ αναφέρονται τα πρακτικά προβλήματα αναφορικά με την εφαρμογή και δύο σταθερές ημερομηνίες προθεσμίες για την εφαρμογή θεωρώ ότι θα βοηθήσουν την όλη διαδικασία εφαρμογή. Θα εξετάσω ποιε προτάσεις ε, θα καταθέσω και σε ό,τι αφορά το θέμα του gold plating για τον κανονικό υπερθεματισμό και την αρχή της επικουρικότητας. Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την συγγητρία για την εξαιρετική έκθεση και προσβλέπω στις περαιτέρω συζητήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Και μια και δεν είναι εδώ η τη από τι άλλε ομάδε, να δώσουμε το λόγο στα μέλη τη Επιτροπή σε περίπτωση που θέλουν το λόγο. Μάλιστα. Ωραία. Θέλει, Αμαλή, να πάρει το λόγο για να συνοψίσει. Ναι, να σα ευχαριστήσω όλου για τις ε, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. Στις 9 Ιουνίου είπαμε ότι ήταν η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και θα διοργανώσουμε το δυνατόν συντομότερο το, την πρώτη συνάντηση των ε, σκιωδών για να υπάρχει μια έκθεση η οποία θα στηρίζεται από όλους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, και τώρα το χρονοδιάγραμμα. 29 Ιουνίου εξεταστή τροπολογιών, 15 Ιουλίου συμβαστικές και ψηφοφορία 16 Ιουλίου. Πολύ ωραία. Και περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση για την πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα. Μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι η καθήλια αρμόδια. Ο Νίκολα Ντάντε είναι συγγητή, αλλά ε, από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ο συγητής, η συγγετρία είναι επίση ε, μέλο τη επική μα επιτροπή και είναι εδώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις πολύ αριθμές τροπολογίες, μεγάλο μέρος των οποίων θα γίνουν δεκτές και θα δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε σημαντικά την ε, γνωμοδότηση, την έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω διότι θεωρώ ότι με αυτές τις τροπολογίες θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση την οποία θα στείλουμε στη συνάδελφο Μπελζίνη Τοζιέ ε, στην Επιτροπή Γιούρη όπου θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ένα σύστημα προστασίας για τα προστασίας γεωγραφικής ένδειξης για μη γεωργικά προϊόντα που θα βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς. Εγώ θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη όλες τις τροπολογίες και να τις συζητήσω και μέσα στις επόμενες ημέρες ε, θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε, να παρουσιάσουμε συμβαστικές τροπολογίες που θα περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι των τροπολογιών που υποβλήθηκαν, θα συμπεριλαμβάνουν την ουσία των στόχων ε, που αποτέλεσαν την αιτία υποβολή αυτών των τροπολογιών. Θέλω να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα, σε ορισμένε τροπολογίε, σε κάποιε προτεραιότητε που χρειάζεται κάποια διευκρίνηση. Ειδικότερα θα ήθελα να ξεκινήσω από τι τροπολογίε 18 του συναδέλφου Πόσπιζιτ που είναι σκιώδη του ΕΛΚΑ και του συναδέλφου Ντε που είναι σκιώδης της ΓΚΟΕ όπου διαφέρεται το γεγονός ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι εθελοντικό. Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω ευθύ εξ αρχή ότι το σύστημα αυτό είναι εθελοντικό. Δηλαδή πουθενά δεν πρόκειται να υποχρεώνουμε να αναφέρεται μια γεωγραφική ένδειξη χωρίς να υπάρξει αίτημα από κάποια ένωση παραγωγών όπως γίνεται για όλα τα γεωργικά προϊόντα, όπου γεωγραφικές ενδείξεις ε, αποτελούν το αντικείμενο αιτήματο από συμπράξεις παραγωγών ή από τοπικούς οργανισμούς, διότι πρόκειται για μια αναγνώριση ε, ε, συλλογικής ονομασίας, ιστορικής σημασίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να είναι υποχρεωτικό, αλλά εθελοντικό εθελοντικό για τους αιτούντε προστασίας για το δικό τους προϊόν. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα περιορίσει το ενδεχόμενο ε, ...καποια άλλη παραγωγή να μπορούν να παράγουν κάτι τέτοιο πέρα της αναγνώρισης της ονομασίας. Από αυτή την άποψη λοιπόν Θεωρώ ότι η νομοθεσία για τα γεωργικά προϊόντα αποτελεί ικανό παράδειγμα και διευκρινίζει αυτό το στοιχείο. Θα το διευκρινίσουμε και εμείς πολύ καθαρά. Διαβεβαιώνω τώρα τον συναδελφό Ποσπιζελ να είναι σαφές από την αρχή ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για υποχρεωτική ε, πιστοποίηση ή ονομασία, αλλά ε, πρόκειται για μια επιπλέον ευκαιρία που προσπαθούμε να προσφέρουμε στους παραγωγούς οι οποίοι παράγουν κάποια προϊόντα τα οποία θέλουν να αναδείξουν ε, μέσω της γεωγραφικής ένδειξης. Τώρα για άλλα ζητήματα, ε, εδώ τώρα κάνω μια διευκρίνηση για πολλές τροπολογίες, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα διότι θα συμβάλλουν ε, στην θετική εικόνα της έκθεσης να σταθώ σε ορισμένες τροπολογίες ειδικότερα στην τροπολογία του συναδέλφου Ντάλτον που δεν βλέπει κάποια θετικά αποτελέσματα για αυτό το ε, ε, αποτελεσματικό σύστημα. Αντιθέτως εγώ πιστεύω ότι το σύστημα αυτό θα βοηθήσει την οικονομία ε, και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης μας όπου παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας και θεωρώ λοιπόν ότι αυτές τις τροπολογίες δεν θα τις δεχτώ. Όπως και επίσης οι τροπολογίες του κ. Ντάλτον και του και συναδέλφου Τρεμπέζιους που ζητούν περαιτέρω ανάλυση και ούτω καθεσής ανάλυση κόστος ωφέλους είναι σαφές ότι θα υπάρξει μια νομοθετική πρόταση θα γίνουν αυτές οι αναλύσεις αλλά εγώ ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι η πρόταση αυτή έχει κάποια ιστορία. Έχουν προηγηθεί αναλύσεις, μελέτες από την Κομισιόν εδώ και πολλά χρόνια. Έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν, ε, είχαμε 136 συμμετοχές από πολλά κράτη-μέλη. Να υπενθυμίσω στον κύριο Ντάλτον 29 ε, συμμετοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο, 28 από τη Γαλλία, 17 από την Ιταλία και Όσοι απαντήσαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρετε, αποτέλεσαν την πλειοψηφία ε, η οποία θεώρησε ότι αυτή η πρόταση ήταν πολύ θετική. Θεωρώ λοιπόν ότι αναλύσεις και βαθύσεις θα γίνουν. Θα γίνουν και όταν θα παρουσιαστεί η νομοθετική πρόταση που ελπίζουμε να εμφανιστεί από την Κομισιόν του χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία μας λένε αντικειμενικά, το λένε τα στοιχεία της Κομισιόν, οι διαβουλεύσεις, ότι η πρόταση αυτή χαίρει τεράστιες αποδοχής από τους παραγωγούς και από τους ενδιαφερομένους. Τέλος, οι τελευταίες τροπολογίες της συναδέλφου Τρεμπέζιος που τείνουν να περιορίσουν το σύστημα αυτό σε εθνικό επίπεδο είναι σαφές ότι εμείς αντιθέτως με αυτή την πρόταση θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση που θα προσφέρει ε, υψηλότερες εγγύσεις σε παραγωγούς ε, πανευρωπαϊκής κάλυψης ε, Οπότε οι τροπολογίες αυτές ε, από εμένα δεν θα γίνουν τουλάχιστον δεκτέ. Ε, κατά τα άλλα, πιστεύω ότι τι επόμενε ημέρες θα καταφέρουμε να συγχωνεύσουμε όλε αυτέ τις τροπολογίε για να καταλήξουμε σε κάποιου συμβιβασμού. Εγώ ζήτησα τους Κιώδη ε, να συναντηθούμε στι 16 Ιουνίου στι Βρυξέλλες, έτσι ώστε να καταλήξουμε συμβαστικέ τροπολογίε που να χαίρουν τι μεγαλύτερε δυνατέ συμφωνίε, δυνατέ συμφωνίε μεταξύ των διαφορών ομάδων. Ε, και στην Επιτροπή αυτή, ώστε 22 Ιουνίου να φτάσουμε ψηφοφορία της γνωμοδότησης ε, και μετά να τα παραδώσουμε όλα στα χέρια της Βρυζίνη η οποία θα μεριμνήσει να ετοιμάσει την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ιουνίου. Ευχαριστούμε Νικόλα, κύριε Σιγητά. Τώρα δίνω το λόγο στον γύρι Προσυπέλ Σκιώδη του ΕΛΚ. Ναι, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα, αν με επιτρέπετε, να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Θεωρώ ότι το έργο του εισηγητού μας, του κυρίου Ντάντη, είναι πάρα πολύ αξιόλογο, εξαιρετικό θα έλεγα. Και συμφωνώ πλήρως μαζί του. Ως και ο εισηγητής του ΕΛΚ σχεδόν συμφωνώ με όλα τα σημεία της γνωμοδότησης. Το θέμα δεν είναι να βρούμε κάποια βαρύγδουπα νομικά μέσα, να δούμε πώς ε, και για μη γεωργικά προϊόντα θα ε, προβλέψουμε παρόμοια προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Σε ό,τι αφορά την εθελοντική βάση, τον εκούσιο χαρακτήρα των ε, ενδείξεων. Αυτό απορρέει και από την πληροφορία που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και καλό θα ήταν να επιμείνουμε σε αυτή την εθελοντική βάση, τον προαιρετικό χαρακτήρα. Και η καταγραφή, σε περίπτωση που γίνεται από τους παραγωγούς, να γίνεται και σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Οπότε, αν έχουμε ευρωπαϊκό μητρό και θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το σύνολο των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα. Αν κατάλαβα καλά, ο εισηγητής είναι δεκτικός απέναντι στις τροπολογίες και τον ευχαριστώ. Θέλουμε την ίδια αρχή που ισχύει για τα γεωργικά προϊόντα σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις να την επεκτείνουμε και στα μη γεωργικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να επενδύσουμε να εφεύρουμε ένα νέο σύστημα, να επινοήσουμε ένα νομικό κατασκεύασμα διαφορετικό. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή. Ευχαριστούμε κύριε Ποσπίσιλ. Ο κύριος Ροσφόρ τώρα από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίες συγχαρητήρια στον Νικόλα. Το κείμενο αυτό είναι εξαιρετικό. Προσφέρει ένα ρεαλιστικό όραμα και συμφωνώ και με τον εθελοντικό χαρακτήρα και το φιλόδοξο χαρακτήρα που πρέπει να το διακατέχει. Πρότεινα λοιπόν ε, κάποιες τροπολογίες. Θεωρώ ότι ο Νικόλα θα μπορέσει να τις ενσωματώσει το κείμενό του. Να κάνω κάποια σχόλια στα γρήγορα. Ναι. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο σήμερα είναι κατακαιρματισμένο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανεπαρκές. Δηλαδή, ενώ πρέπει να παραμένουμε ρεαλιστές ε, επιβάλλεται το σύστημα αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων να είναι ενοποιημένο να είναι ευανάγνωστο να μπορεί να αναγνωριστεί ως παρομοιότυπο για τις διάφορες προελεύσεις στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή εξορισμού ευνοεί την ποιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω θα πρέπει στις σημερινές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς θα πρέπει να παρέχει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Κάθε φορά λοιπόν που προτείνουμε οτιδήποτε κάποια γεωγραφική ένδειξη ε, που ε, βελτιώνει την ποιότητα αυτό αποτελεί και κίνητρο για, την, ε, για τους παραγωγούς να παίξουν το χαρτί της ποιότητας και σε μη γεωργικά προϊόντα. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα να επισημάνω ε, το σύστημα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβάλλει κάποιο προστατευτισμό, ότι προορίζεται μόνο για Ευρωπαίους που καταναλώνουν πράγματα μεταξύ τους. Θα εξυπηρετήσει και τις αγορές τρίτων χωρών. Θα δίνει τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο παραγωγό να αποκτήσει νέες αγορές πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόμενος μόνο σε αυτές ε, τις γεωγραφικές ενδείξεις που θα αποτελούν πλέον πλεονέκτημα για τις εξαγωγές. Αν με επιτρέπετε άλλα δύο-τρία σχόλια όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων όταν θα ξανοιχτούν ε, και όταν θα... η Κομισιόν θα κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εργαζόμαστε. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να τις επιβαρύνει με διατυπώσεις. Ε, θα πρέπει να είναι κάτι απλό, εναρμονισμένο. Εναρμονισμένο με ένα αλλά απλό. Επίσης, ε, στην παρουσίαση σας πριν λίγα λεπτά αναφερθήκατε σε κάτι άλλο. Οι όμιλοι παραγωγών, οι ενώσεις, οι οργανισμοί, οι προξενικοί οργανισμοί, οι, ε, τοπικοί, οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια γεωγραφική ένδειξη για τα μη γεωργικά τους προϊόντα. Είναι κάτι που θα χρησιμεύσει όλους. Και τέλος ε, να πω ότι ε, κοιτώντας όλα αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να ξεχνάμε την πτυχή της ενημέρωσης του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει την προέλευση της γεωγραφικής αυτής ενδείξης. Πρέπει να ξέρουμε ότι σήμερα Υπάρχει κάποια σύγχυση πολλές φορές μεταξύ εμπορικών μαρκών, γεωγραφικών ενδείξεων και γεωρισμένα προϊόντα που έρχονται από την Ιταλία και που αρχικά, από την Ιταλία αρχικά είναι ιταλικής προέλευσης ε, πρέπει να είναι πιο σαφείς οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή ώστε αυτός να μπορεί να αναγνωρίζει πραγματικά τι είναι η γεωγραφική ένδειξη που έχει μια εμπορική αξία αλλά που δεν είναι εμπορική μάρκα. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Νικόλα Ντάντη και να υπενθυμίσω ότι είμαστε στη διάθεσή του για να συνεργαστούμε ε, για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες το συντομότερο. Ευχαριστούμε Ρομπεροσφόρ, δίνω το λόγο εδώ στη Βυζινή Ρουζιά. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ω εισηγήτρια τη έκθεση ε, τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, ευχαριστώ τον Νικόλα για την πολύ αξιόλογη γνωμοδότηση που συνέταξε, αλλά και την αγαστή συνεργασία που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και που ευελπιστώ θα συνεχιστεί ε, μέχρι τις ψηφοφορίες και στην ΙΜΚΟ και στη Γιούρη. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας μας και τη στήριξαν. Συμφωνώ ότι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας ε, ε, τη τοπική παραγωγή ανταποκρίνεται σε αιτήματα χνηλασιμότητας ε, και αυθεντικότητα των ε, καταναλωτών και θα ωφελήσει και τι επιχειρήσει αλλά και τι περιφέρειες. Ευχαριστώ τον Νίκολα που τόνισε τον προαιρετικό χαρακτήρα αυτών των μέτρων. Γιατί πάνω απ' όλα θα πρέπει να εξυπηρετούν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει να σταθούν στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν την παραγωγή τους. Και όπως γίνεται με τις γεωγραφικές ενδείξεις στα γεωργικά προϊόντα, θα μπορούσαμε αυτό το σύστημα να το χρησιμοποιήσουμε και τα μη γεωργικά προϊόντα. Γιατί όπως είπε ο Ρομπέρο Φόρ, αυτή η αναγνώριση της ποιότητας της γεωγραφικής ένδειξης είναι σημαντικός μοχλός για την κατάκτηση αγορών εξαγωγών. Έχουν φανεί τα πλεονεκτήματα για τα γεωργικά προϊόντα, θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε μη γεωργικά προϊόντα, εφόσον ε, το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων το χρησιμοποιήσουμε και σε αυτά σε ό,τι αφορά τις μελέτες, τις έρευνες ε, και τα πορίσματα, θα ήθελα να υπενθυμίσω την ιδιαίτερη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν και αρκετά εμπεριστατωμένη και ογκώδης το 2013 που αναλύει διάφορες προτάσεις και καταλήγει σε συστάσεις. Ήταν ε, πολύτιμη η ε, συμβολή αυτής της μελέτης. Και επίσης είχαμε και την διαβούλευση, τη γενική που ολοκληρώθηκε αυτή τη βδομάδα με συμμετοχή ε, ε, των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων που τάσσονται υπέρ του συστήματος. Μερικοί Γάλλοι ε, έχουν ένα πρόβλημα και εξέφεσαν τη λύπη τους για το δεν για το εθνικό επίπεδο. Μάλιστα είχαμε τώρα πρόσφατα ένα εθνικό ζήτημα και μάλιστα προστασία εθνική για τι γεωγραφικέ οπότε το θέμα θεωρείται λήξαν. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πρέπει να αναζητηθεί η λύση. Γιατί η ευρωπαϊκή εναρμόνιση θα είναι μοχλό απλούστευση, γιατί θα έχουμε καλύτερο επίπεδο προστασία στο σύνολο τη ευρωπαϊκή επικράτεια και μία ενιαία διατύπωση για τι 28 χώρε μέλη. Επιθυμητή απλούστευση για τι επιχειρήσει και δι τι μικρομεσαίε. Και εδώ στηριζόμαστε στι ρυθμίσει που ίσχυσαν για τα γεωργικά προϊόντα και έχουμε τον ειδικό ρόλο του OSME γιατί σίγουρα η συνύπαρξη με τα εμπορικά σήματα είναι σημαντικό θέμα για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Ευχαριστώ και πάλι θερμά τον Νικόλα Ντάντη για την αξιόλογη γνωμοδότησή του και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ Βαλερή. Βι... Βυρζινή μάλλον. Η Βαλερή τώρα θα μιλήσει. Ε, η Βαλερή Νταβινιό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή μάλλον ο Βαλερή Νταβινιό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε το θέμα αυτό, η κυρία Κέννη και εδώ, οι συνάδελφοι. Παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα αυτό πάρα πολύ ε, επισταμένος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σα ευχαριστώ πάρα πολυ επισταμενος δεν θελω να μακρηγορησω Σα ευχαριστω παρα πολυ για τι χρήσιμε παρεμβάσει σα και ασφαλώ και τον εισηγητή για το σημαντικό αυτό έργο του. Νομίζω ότι πολλά από τα σημαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο αυτό έχουν αναφερθεί σε λούσια βάση, ένα εργαλείο που θα ειδετεθεί σε όλους όσους ε, θέλουν να αποφεληθούν από αυτό. Πρόκειται για θέματα ποιότητας, για θέματα ενημέρωσης του καταναλωτή και θα πρέπει να είναι ελαφρύ, αποτελεσματικό προκειμένου να μπορέσει να αποδώσει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις. Προσβλέπουμε λοιπόν στο τελικό αποτέλεσμα των διαβουλεύσεών σας ε, μετά από τις απόψεις και των υπόλοιπων επιτροπών και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει σημαντικά στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό. Πριν από λίγες ημέρες, όπως αναφέρθηκε, δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα της ε, δημόσιας διαβούλευσης, μία σύνοψη των αποτελεσμάτων. Χρήσιμο λοιπόν και ωφέλιμο αν θέλετε να διαβάσετε. Να σας ευχαριστήσω επίσης για την πληροφόρηση ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία στην Γαλλία, γιατί προφανώ πρόκειται για ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε στενά, η πρακτική εμπειρία σε εθνικό επίπεδο είναι χρήσιμη. Και μετά, αφού έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία αυτά, θα περάσουμε στο επόμενο βήμα. Και είμαστε φυσικά στη διάθεσή σας για συζήτηση όποτε χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο σκιώδης των Πρασίνων, ο κ. Σόλτας κατέφτασε. Ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι και αποτελεσματικοί σήμερα το πρωί. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεση. Η Επιτροπή μας δεν ε, ασχολείται μόνο με την εσωτερική αγορά, αλλά προασπίζει και τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ω εκ του πρέπει να τονίσουμε ότι η γεωγραφική ένδειξη είναι σημαντικό ζήτημα και για τη διαφάνεια και ασφαλώς βοηθά τον καταναλωτή στην επιλογή των προϊόντων του. Για την καλύτερη λοιπόν ενημέρωση. Οι πράσινοι κατέθεσαν δύο τροπολογίες με τις οποίες θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η γεωγραφική ένδειξη δεν, εγκυάται δεν εγγυάται την ανεχνευσιμότητα ασφαλώ, αλλά την διευκολύνει για την καλύτερη ανιχνευσιμότητα θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν και η νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων στην αγορά να βελτιωθεί. Και αυτά είναι σημαντικά για την προάσπιση των συμφέροντων του καταναλωτή και θα πρέπει να λεφτεί υπόψη ασφαλώ και η συμφωνία TTIP. Αν η Ευρώπη έχει και ψηφίσει προδιαγραφές και κοιτάξει για την γεωγραφική ένδειξη, τότε ασφαλώ. αυτό θα πρέπει να διαδηματίσει ρόλο και στην συμφωνία TTIP, γιατί και τα κράτη-μέλη του τι θα πρέπει να αναλάβουν αυτές, να αποδεχτούν αυτές τις ε, διατάξεις. Ο Νίκλα Ντάντε, αν θέλει να συνοψίσει. Να ευχαριστήσω για τη συζήτηση, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα καταφέρουμε να παρουσιάσουμε μια ομάδα από συμβιβαστικές τροπολογίες που θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις προτάσεις σας οι περισσότερες από τις οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση που είπαμε, ένα ευρωπαϊκό και όχι εθνικό σύστημα απλό που να προσφέρει όμως τη δυνατότητα σε πολλούς παραγωγούς ποιότητας να έχουν ε, σήματα τα οποία όπως ε, και στο γεωργικό τομέα μπαίνει κάποιος από εμάς στο σούπερ μάρκετ χωρίς να γνωρίζει τίποτα από κρασιά αλλά βλέπει τη γεωγραφική ένδειξη, την ευρωπαϊκή ονομασία αυτή ως σύμβολο ποιότητας. Ελπίζουμε να γίνει το ίδιο και για τα μη γεωργικά προϊόντα της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, ε, ε, κατά την άποψή μου, όλες οι τροποποίησεις, ε, όλες οι τροπολογίες που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν προσδεκτής και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια εκθέση που θα δώσει μια μεγάλη όθηση στην Κομισιόν του χρόνου από την, από την Επιτροπή Γιούρη φυσικά για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε Νικόλα. Χρονοδιάγραμμα θα ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ 22 και 23 Ιουνίου. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα Γερμανών επισκεπτών που βρίσκονται μαζί μας εδώ και λίγη ώρα και που ε, επισκέπτεται το βουλευτή Καλώς ορίσατε. Κλείνουμε εδώ τη συνεδρίαση γιατί δεν έχουμε τίποτα από τα διάφορα. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις... Ε, Α, Εύελιν, έχετε το λόγο. Έχω ένα θέμα να θέσω στον διάφορα. Χθες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώθηκε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για τα 10 έτη προστασίας του Ευρωπαίου καταναλωτή. Ήταν πολύ καλή λοιπόν η εκδήλωση και με συζήτηση, μετά από συζήτηση των εκπροσώπων των κέντρων καταναλωτών, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αγνοούν πολλοί συνάδελφοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να σκεφτούμε σε μία από τις μεραδικές συνεδριάσεις πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τους βουλευτές για αυτό το πάρα πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο εργαλείο. Και άμα όταν έχουν πρόβλημα οι καταναλωτές να διαβιβάζονται, να τους παραπέμπουν στα κέντρα αυτά. Γιατί πραγματικά η ενημέρωση εκεί είναι πολύ υψηλή ποιότητα και θα πρέπει ω καταναλωτέ να τα γνωρίζουμε. Thank you, Evelyn. Σα ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Να το συζητήσουμε στη συνάντηση των συντονιστών. Στι 22 και 23 Ιουνίου είναι η επόμενη συνεδρίαση. Σα ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.